Καλή σας μέρα. Ξεκινούμε λοιπόν τη συνεδρίασή μας. Δεν βλέπω να υπάρχουν παρατηρήσεις και σχόλια επί τη προτινόμενης ημερησίας διατάξεως, επομένως θεωρείται εγκεκριμένη. Δεν έχω λάβει ερωτήσεις για την Επιτροπή. Δεν έχω και ανακοινώσεις. Επομένως... Avez reçu dans votre dossier Έχετε στα έγγραφά σας ε, τις ε, συστάσεις καθώς επίσης και τις αποφάσεις που ελήφθησαν από τη Συνεδρία των συντονιστών της 7ης ε, Νοεμβρίου 2011. Εάν έχετε σχόλια για παρατηρήσεις από αυτόν, παρακαλώ να το πείτε στην γραμματεία, διαφορετικά θα εγκριθούν τα πρακτικά αυτά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να πάρει το λόγο, έχει κάποιες ανακοινώσεις να μας κάνει. Όχι από ό,τι φαίνεται. Επομένως, περνούμε εις ε, την κανονική ημερήσια διάταξη, σημείο 6 λοιπόν. Ε, ε, προβλέπεται λοιπόν βάσει του σημείου 6 ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις γενικευμένες προτιμήσεις. Η κυρία Στρίφλερ έχει το λόγο, είναι η εισηγήτριά μας για το σύστημα γενικευμένων δεσμολογικών προτιμήσεων ο κανονισμός του 2008 για το ε, θέμα ε, αυτό αυτό ε, υπέρ των χωρών, ε, των αναπτυσσόμενων χωρών ε, εκπνέει το 2013 και επομένως θα πρέπει να ανανεωθεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημοσιεύσει μία πρόταση η οποία πρέπει να επικαιροποιηθεί. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα το οποίο θα πρέπει να ειδωθεί βάσει της θέσης σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας και η Επιτροπή Ίντα ξέρετε ότι είναι υπεύθυνη επί της ουσίας. Κυρία Στρίφλερ, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πριν ξεκινήσω θα ήθελα να σας δώσω και μία σημαντική πληροφορία. Η κυρία Εύα Ζολή σήμερα γιορτάζει τα γενέθλιά της. Παρακαλώ να χειροκροτήσουμε όλοι. Δεν μπορούσα να το ξεχάσω αυτό. Είναι σημαντική η περίσταση. Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι γεγονός ότι πρόκειται για θέμα πολύ σημαντικό. Θα προσπαθήσω να μην μακρηγορήσω, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να σας δώσω κάποιες εξηγήσει. Ε, το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων γνωρίζετε ότι είναι στρατηγικό εργαλείο της, πολιτικής, ε, της αναπτυξιακής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, προτίθεται να στηρίξει τις προσπάθειες ανάπτυξης των αναπτυσσόμενων χωρών δίνοντας ταυτόχρονα προτεραιότητα εις ε, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ε, αηφόρο ανάπτυξη. Έχουμε το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων κλασικό, καθώς επίσης και το ειδικό σύστημα το οποίο δίνει σε 176 χώρες ε, η προ, προτιμησιακό καθεστώς πρόσβαση στην αγορά. Βεβαίως στηρίζουμε με το SPG Plus ε, την καλή διακυβέρνηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, όλα, σε όλα αυτά τα ονομάζουμε TSA. Η νέα πρόταση που μας έχει υποβληθεί ε, τροποποιεί κατά, κατά ε, πολύ τις ε, καταστάσεις όσον αφορά τις αναπτυσσόμενες χώρες και βεβαίως στοχεύει κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, τις αναπτυσσόμενες χώρες οι οποίες έχουν περισσότερη ανάγκη, δηλαδή τις φτωχές και πολύ φτωχές χώρες. Μία από τις πιο σημαντικές αλλαγές οπωσδήποτε είναι η μείωση των χωρών ε, που ε, εμπίπτουν στο σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων. Δηλαδή από 176 χώρες ε, και εδάφη περνάμε σε περίπου 80 χώρες που ωφελούνται από το σύστημα. Τρεις, χώρ, τρεις ομάδες χωρών στόχων δεν θα στοχεύονται πλέον από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ναι, αυτές ε, οι οποίες ε, έχουν ε, ειδικό καθεστώς, οι χώρες αυτές οι οποίες αποτελούν είτε υπερπόντια διαμερίσματα χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε της Αυστραλίας, καθώς επίσης και τρίτη ομάδα, οι χώρες οι οποίες έχουν περάσει σε ένα επίπεδο εισοδημάτων αρκετά υψηλό. Ε, οι δύο πρώτες ε, ε, χώρες ενδεχομένως δεν θα μας δημιουργήσουν ιδιαίτερο πρόβλημα. Στην τρίτη κατηγορία χώρων όμως θα έχουμε πρόβλημα. Ε, όσον αφορά το θέμα της χρήσης ε, του δίκτυ της Παγκόσμιας Τράπεζας θεωρώ ότι ε, το να θεωρήσουμε μοναδική προϋπόθεση το κατακεφαλήν εισόδημα θα μπορούσε να, είναι, να καταλήξει σε ένα σύστημα κυρωτικό για τις μικρές χώρες οι οποίες σε ορισμένες περιοχές αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο πρόβλημα φτώχειας. Ε, γι' αυτό λοιπόν, παρότι συμφωνώ σε γενικές γραμμές με το κριτήριο αυτό, θεωρώ ότι παρόλα αυτά παρουσιάζει κάποια ασθενή σημεία τα οποία θα πρέπει να μελετηθούν. Θα ήθελα επίσης να υπενθυμίσω ότι τα τελευταία χρόνια ήταν ταραχώδης η ακαδημαϊκή συζήτηση και η πολιτική ε, εν μέρη συζήτηση σχετικά ε, με το κατά πόσον οι οικονομικοί δείκτες μπορούν να αποτελέσουν στοιχείο μέτρησης της αηφορίας επίσης ε, ε, και ε, ειδικότερα της κοινωνικής ή περιβαλλοντικής αηφορίας. Ε, ας πούμε, ο, πρόεδρο, ο, ο, ο καθηγητής Στίγκλιτς, ο οποίος ήταν Νόμπελ Οικονομίας, πρόσφατα προείδευσε ομάδας εργασίας του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, όπου θεωρήθηκε ότι θα πρέπει να μπουν και άλλοι δείκτες, όπως είναι η κοινωνική ευημερία και άλλοι. Ε, πιστεύουμε λοιπόν ότι θα πρέπει να δούμε ε, ε, επίσης ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι εξειδικευμένα μπορούν να μας δώσουν σωστές πληροφορίες, να δούμε, να έχουμε κάποια σημεία αναφορά όσον αφορά το πρόγραμμα αυτό, καθώς επίσης και τη διασύνδεση του προγράμματος αυτού και των στόχων με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όσον αφορά τώρα τις διεθνείς, τις διεθνείς συμφωνίες οι οποίες θα πρέπει να να επικυρωθούν. Είμαι σύμφωνη με, με τον κατάλογο αυτών των 27 χωρών, άρα 27 συμφωνιών. Οπωσδήποτε θα πρέπει να βελτιώσουμε περαιτέρω τις υπάρχουσες συμφωνίες πριν ε, προσπαθήσουμε να διευρύνουμε με παράλογο τρόπο ή μη ρεαλιστικό τρόπο τις ε, ε, συμφωνίες αυτές. Επίσης, χώρες όπως το Περού, η Κολομβία ή άλλες χώρες τη Κεντρικής Αμερικής, οι οποίες έχουν ε, ειδική διμερή συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε χώρες οι οποίες έχουν περάσει στην παραπάνω κατηγορία των όχι ε, πολύ φτωχών χωρών, που πλέον δεν εμπίπτουν στο σύστημα γενικευμένων ε, τιμήσεων, θα πρέπει να μα απασχολήσουν ιδιαίτερα. Επίσης, ε, χρειαζόμαστε ορθές πρακτικές όσον αφορά ε, την παράνομη εκροή κεφαλαίων, την ε, φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή, την σωστή οικονομική διακυβέρνηση και την δημοσιονομική εξυγίανση. Οπωσδήποτε όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία θα πρέπει να μας απασχολήσουν στα πλαίσια της επικαιροποίησης του συστήματος γενικευμένων προετοιμήσεων. Οπωσδήποτε επίσης θέλουμε να ευχαριστήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για την καλή συνεργασία που είχαμε και βεβαίως παραμένω στη διάθεσή σας για την περαιτέρω συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κέλλερ έχει το λόγο. Thank you. Uh, and thank you very much. Uh, σας ευχαριστώ κυρία Στίφλερ για την έκθεσή σα. Εμεί οι βλέπουμε θετικά στοιχεία στην πρόταση της Κομισιόν Όπω ότι διατηρούνται τα τρία σχέδια, ότι υπάρχουν ε, διαγραφές ορισμένων πιο πλουσίων υπερπόντιων ε, εδαφών και ότι ορισμένες χώρες μπορούν τη στιγμή να ζητήσουν ε, το, να συμμετάσχουν στο σχέδιο GSP συν. Υπάρχουν υποθετικά στοιχεία, έχουμε και κάποιες ανησυχίες όμως. Η κυρία μας ανησυχία είναι ότι αν χρησιμοποιηθεί το κριτήριο του εισοδήματος, που είναι η μόνη μέθοδος που προτείνεται, το μόνο κριτήριο, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί και το μέσο του GSP ως μέσο ανάπτυξης. Το αριθμός των δικαιούχων θα μειωθεί από 176 σε 80 περίπου. Πάρα πολύ σοβαρή μείωση δηλαδή. Το θέμα είναι κατά πόσον αυτή η τόσο δραστική μείωση θα ωφελήσει τις υπόλοιπες χώρες. Δεν ανησυχούμε βέβαια τόσο πολύ για την διαγραφή των 35 υπερπαντίων διαμερισμάτων των πλουσίων χωρών. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν ε, κάποιες χώρες με σχετικά ψηλό εισόδημα που δεν έχουμε τη δυνατότητα όμως για συνθήκες ελευθέρων συναλλαγών ή εμπόριο μέσα στα πλαίσια του, του, ε, της, ε, διεθνούς, ε, του Διεθνούς Οργανισμού Εμπορίου και συμπεριλαμβάνουν και κάποιες φτωχές χώρες, η Ναμίβια, το Εκουαντόρ και το Αζερβαϊτζάν. Και άμα πάρουμε τις προατιμήσεις από αυτού του τύπου τις χώρες, θα τις πιώσουμε σε συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών ελεύθερε συναλλαγέ, όμω είναι κάτι που θα πρέπει να κάνει κανένα ελεύθερα, όχι επειδή πιέζεται να το κάνει. Η εκτίμηση επιπτώσεων της Κομισιόν καταδεικνύει επίσης ότι το θέμα του ποιος θα ωφεληθεί εάν αφαιρεθούν όλες αυτές οι χώρες από το σχέδιο δεν θα είναι οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες τελικά. οι Παγκλατές παραδείγματος χάρη θα χάσει 25 εκατομμύρια περίπου με τη μεταρρύθμιση αυτή. Και φαίνεται ότι όσο πιο πολλά ωφέλη υπάρχουν στις χώρες του ΩΣΑ, τόσο λιγότερο ωφελούνται οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Δεν φαίνεται να συμβαίνει αυτό, σύμφωνα με την εκτίμηση της ίδιας Κομισιόν. Τέλος, το θέμα των κριτηρίων. Συμφωνώ με αυτό που προτείνετε, να έχουμε τον δίκτυο ανθρώπινης εξέλιξης στο αγγλικό κείμενο της Τροπολικής παρελθόν 2 λέει θα πρέπει να ληφθεί επίσης υπόψη και οποιοδήποτε άλλο σημαντικό κριτήριο μεταξύ των οποίων και η ανταγωνιστικότητα. Δεν ξέρω. Αυτό είναι θέμα τώρα του κειμένου, μεταφράσει του κειμένου. Εσείς δεν το αναφέρατε αυτό, μήπως θα πρέπει να το εξάσουμε αυτό, να μας το διευκρινίσετε κατά δυνατόν. Το ε, παράθυρο ευκαιρία για την προώθηση της περιφερειακής ολοκληρωσής είναι επίσης πολύ σημαντικό, το κάνει στην Αφρική. Γιατί μια χώρα έχει αυτό το σχέδιο στο οποίο έχει ενταχθεί η άλλη το άλλο και θα ήταν καλό λοιπόν να κάνουμε κάτι το πιο συγκεντρωμένο, μια πιο περιφερειακή προσέγγιση. Τελευταίο ερώτημα αφορά την τροπολογία βαριθμών 1. Δεν κατανοούμε ακριβώ τι εννοείται η ταξινόμηση σας ενδιαφέρει ή θέλετε να συμπεριλάβετε και τις δικαιούχες χώρες που ακόμα δεν ωφελούνται, αλλά θα μπορούσαν να ωφεληθούν. Ευχαριστώ πολύ ευχαριστώ. Η κυρία Ότ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα κι εγώ να χαιρετήσω το σχέδιο γνωμοδότησης της ηγετρίας και συμφωνώ <coughs> με αυτά τα οποία είπε προλαλήσασα. Δηλαδή, ότι θα πρέπει τον δίκτυο ανθρώπινης ανάπτυξης να τον συμπεριλάβουμε εδώ όχι μόνο το GNI. Νομίζω ότι έχουμε πρόβλημα με τις χώρες μέσης σε ανώτερης ανάπτυξης. Κάποιες χώρες έχουν βρεθεί ακόμη και όταν εξαρτώνται από έναν μόνο τομέα. Αλλά η ποικιλία των χωρών και ο αριθμός των χωρών που βρίσκονται σε αυτή την κατηγορία είναι αρκετά σημαντικός παρά το γεγονό ότι κάποιε από αυτέ έχουν αποκλειστεί, διότι ίσω έχουν υπογράψει συμφωνίε ελεύθερη πορεία και έχουν ούτω ή άλλως με άλλο τρόπο τα συστήματα γενικευμένες προτιμής, υπάρχουν και άλλες χώρες που κινδυνεύουν παρόλα αυτά να χάσουν εντελώς, διότι είναι σε μία ενδιάμεση κατηγορία ανάμεσα στις διάφορες θέσεις που αναφέρονται εδώ. Και ιδιαίτερος η αλλως με αλλο τροπο τα συστηματα γενικής προτιμης υπαρχουν και αλλες χωρες που κινδυνευουν παρολα αυτα να χασουν εντελως διοτι ειναι σε μια ενδιαμεση κατηγορια αναμεσα στις διαφορες θεσεις που αναφερονται εδω και ιδιαιτερος η μποτσουανα και η Ναμιμπία έχουν πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση να αντιμετωπίσουν εξαιτία των ελληνικών συμφώνιων που υπάρχουν με την Νότια Αφρική. Θα πρέπει λοιπόν αυτές τις χώρες μεσαίου εισοδήματος, το λάβουμε υπόψη, και οι δείκτες επίσης της ανθρώπινης ανάπτυξης και εξέλιξης νομίζω ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στα πλαίσια του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων. Εάν λοιπόν θεσπίσουμε το κριτήριο αυτό του δίκτυα ανθρώπινης εξέλιξης για αυτές τις χώρες, πιστεύω ότι θα κάνουμε κάτι πολύ σημαντικό. Ποιος είναι ο στόχος του να έχουμε αυτό το σύστημα. Να βοηθήσουμε την ανάπτυξη των χωρών αυτών. Και το GSP, το σύστημα αυτό το SIN, είναι ένα ισχυρό μέσο για να προωθήσουμε την αηφόρο ανάπτυξη. Χαιρετίζω λοιπόν αυτό το οποίο αναφέρεται στην πρόταση που θα πρέπει να γίνει αυτό το GSP συν πιο σημαντικό. Διερωτώ μου όμως ότι αν δεν θα έπρεπε προς αυτήν την κατεύθυνση να είμαστε κάπως πιο φιλόδοξοι. Διότι όσο έχουν τα πράγματα, μόνο δύο χώρες εδώ ε, είναι ε, επιλέξιμες για να μπουν σε αυτό το σύστημα. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να αυξήσουμε το ποσοστό από 2 σε 2,5-3% ώστε να μπορέσουν να εισαχθούν σε αυτό το σύστημα το ΣΥΝ και άλλε χώρε και να μπορέσει να γίνει αυτό το σύστημα πιο ελκυστικό. Διότι έτσι μόνο νομίζω ότι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και τα προβλήματα της τήρησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλα κοινωνικού τύπου κριτήρια που θα πρέπει να βάλουν υπόψη. Επίσης, θα, τον τρόπο θα υπάρχει δυνατότητα να προσθεθούν και συμπληρωματικά προϊόντα στο σύστημα γενικευμένων προεκτιμήσεων ΣΥΝ. Πιστεύω ότι θα πρέπει να μελετηθεί περαιτέρω το πρόβλημα ώστε να μην χάσουν επιδημένες χώρες αλλά να μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες και να στοχοποιήσουμε περισσότερο χώρο. Θα ήθελα να είναι πιο φιλόδοξο σχέδιο της Επιτροπής. Επίσης, η Επιτροπή άλλαξε κάπως τη διατύπωση όσον αφορά τα κριτήρια και λέει ότι θα πρέπει να αποφευθούν οι αθέμητες προοπτικές ανταγωνισμού, κυρίως αυτές που αφορούν και την ε, παροχή πρώτων υλών. Θα ήθελα να μας πει τι εννοεί και γιατί περιλαμβάνει εδώ και τις πρώτες ύλες η Επιτροπή. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Νόισερ έχει το λόγο. Είναι πάρα πολύ φορτωμένο το πρόβλημα. Παρακαλώ κύριε Νόισερ να είστε σύντομος. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρο και ευχαριστώ και την κυρία Σνίφρα για την έκθεσή της. Θεωρώ ότι θα πρέπει να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στο τι σημαίνει ΓΣΠ. Το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων είναι ένα μέσο της ε, συνεργασίας για την ανάπτυξη και χαιρετώ το γεγονός ότι τα κριτήρια ε, βάσει των οποίων δίνεται η ενίσχυση διευρύνονται. Οπωσδήποτε θέλουμε την προστασία των ανθρωπινών δικαιωμάτων, Οπωσδήποτε θέλουμε σαφή κριτήρια για μια αηφόρο ανάπτυξη. Ο στόχος των ε, ΓΣΠ θα πρέπει να είναι ότι θα πρέπει να ωφελούν τους πιο φτωχούς των πιο φτωχών χωρών. Δεν έχω μεγάλη κατανόηση αν ισχυρέ χώρε όπως η Ινδία και η Κίνα εξακολουθούν να συμπεριλάβονται στον κατάλογο αυτό. Θα πρέπει να αποστείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ακριβώς ε, η Ινδία που έχει τόσο φιλόδοξο πρόγραμμα διαστημικών ερευνών προωθήσει, πώς θα εξηγήσουμε στο φορολογούμενό μας ότι ενισχύεται από μας. Θα πρέπει στις χώρες αυτές να μειωθεί ο όγκος ενισχύσεων σίγουρα. Τελευταίο σημείο, η αναφορά για μια λογική πολιτική φορολόγησης και η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Αυτά είναι πάρα πολύ σωματικά κριτήρια πάνω στα οποία θα πρέπει να στρέψουμε και εμείς την προσοχή μας. Ευχαριστώ πολύ. Merci. Ευχαριστώ. Thank you, Mrs. Chairman. Um... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για όλα τα σχόλιά σας. Σίγουρα ήταν πολύ εύστοχες οι ερωτήσεις που κάνετε κυρίες και κύριοι. Είναι πολύ πολύπλοκο το θέμα. Γι' αυτό το λόγο, κοιτάξτε με παρακαλώ, γι' αυτό κάναμε αυτό το ενημερωτικό έγγραφο, το οποίο ελπίζουμε ότι θα μπορέσει να σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα αυτό το πολύπλοκο θέμα όσο προχωρούν οι συζητήσεις. Και θα γίνει η ενημέρωση αυτής της ε, ε πληροφόρησης βάση των τι ε, που αναφέρατε. Γι' αυτό σας ευχαριστώ που κάνετε αυτό που κάνετε. Σας ευχαριστώ για την ε, προσωρινή έκθεση της κυρίας Τρίφρα και για την υποστήριξη των ε, ιδεών που παρουσιάζουμε, δηλαδή δεν είμαστε πιο γενναίο στα πλαίσια με αυτό το στιγμή. Θα ήθελα, λαμβάνοντα υπόψη αυτά τα οποία είπατε, να μπορέσω να σας απαντήσω λέγοντας ότι να μην ε, σας οδηγούν σε λάθη αυτά που βλέπετε με τους αριθμούς. Λέτε ότι πρόκειται για πάρα πολύ η ουσιαστική αλλαγή, διότι πάμε 176 σε 80 και κάτι χώρος. Αν κοιτάξετε λίγο ότι ποιοι είναι αυτοί οι δικαιούχοι και ποιοι θα χάσουν την πρόσβαση σε αυτό το σύστημα, μιλούμε μόνο για χώρες μέσου ως ανώτερου μόνο για 12 χώρες μόνο. Όλες οι άλλες ή με άλλο τρόπο θα έχουν πρόσβαση σε διμερείς συμφωνίες ή πρόσβαση στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή θα μπουν στην κατηγορία των υψηλών εισοδημάτων και θα συμφωνήσετε φαντάζομαι μαζί μου ότι εδώ δεν είναι η ομάδα στόχος την οποία θέλουμε να βοηθήσουμε όπως η Σαουδική Αραβία, το Αμάν, το Κατάρ και το Μπρουνέι. Αυτό είναι πολύ σημαντική πρώτη παρατήρηση. Δεύτερη, η ε, μελέτη εκτίμηση έδειξε ότι οι λιγότερο αναπτυγμένε χώρες φαίνεται ότι βρίσκονται εδώ χωρίς καμία αλλαγή δεδομένου ότι αν δεν κάνουμε κάτι με το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων θα χάσουν. Ή λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε κάτι ώστε να αυξήσουμε τις ε, οι εισαγωγέ, οι εξαγωγές και προσοδές σε εμά ή θα χάσουν πολλά εκατομμύρια. Το πρώτο λοιπόν πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να εφαρμόσουμε αυτό το σύστημα σε αυτούς που έχουν περισσότερη ανάγκη κάνοντας, αφήνοντα την κατάσταση όσο έχει ώστε να μην χάσουν αυτέ οι χώρε. Έτσι θα πρέπει να εννοήσετε αυτές τι ε, αλλαγές. Περισσότερε, λιγότερο ανεπτυγμένε χώρε θα υποφεληθούν μόνο με ένα ε, παράδειγμα, το οποίο, μια εξαίρεση όπως αναφέρεται το Μπαγκλαντές. Και αυτό έχει σχέση με ένα άλλο στοιχείο το οποίο αναφέρεται. Έχει σχέση με το gsp Συν. Εάν θέλουμε να αναπτύξουμε αυτό το σύστημα και να το εφαρμόσουμε σε χώρες όπως το Πακιστάν ή οι Φιλιππίνες, το Πακιστάν και οι Φιλιππίνες θα είναι σε μεγαλύτερο ανταγωνισμό με τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες όπως το Μπαγκλαντές. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι στην Ευρώπη δεν μπορούν οι εισαγωγέ και εξαγωγέ να είναι ανταγωνιστικέ. Αν δεν ακολουθήσουμε σωστά λοιπόν το σύστημα που θέλουμε να εφαρμόσουμε, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τίποτε το σωστό. Γι' αυτό μειώσαμε τον αριθμό των δικαιούχων. Ευχαριστώ. Έχετε το λόγο κυρία Στίφλα για να ολοκληρώσετε πάρα πολύ σύντομα. Δύο λεπτά. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά τα οποία είπαν οι συνάδελφοι. Μία διευκρίνηση για την κυρία Κέλλερ μόνο. Εγώ δεν ξέρω αν έγινε, ε, έγινε μετάφραση στα αγγλικά. Δεν μπορώ να διαβάσω αγγλικά. Στο παρατροπολογία 2 μιλώ για κάτι γενικό. Εάν θέλετε μπορούμε να το συζητήσουμε αργότερα, αλλά η βασική τροπολογία είναι η 1. Δεν ξέρω αν μπορέσατε να καταλάβετε αυτά τα οποία είπε, θα τα πούμε αργότερα αν θέλετε. Υπενθυμίζω, η νομοδότηση θα ψηφιστεί 24 Ιανουαρίου και μέχρι τις 6 Ιανουαρίου έχετε προθεσμία κατάθεση τροπολογιών ως τις 5 ώρα το απόγευμα. Και τώρα θα περάσουμε στο επόμενο θέμα, το σημείο 7 της ημερήσιας διάταξης, παρουσίαση του προγράμματος εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της επιχειρησιακής στρατηγικής για το 2012 της Γενικής Διάθεσης ΕΚΟ από την ε, Επίτροπο κυρία Τζόρτζεβα, η οποία θα μπει σε ένα λεπτό στην αίθουσα. Donc, να σας καλωσορίσω, κυρία Τζόρτζεβα. Θα μας παρουσιάσει, κυρία Τζόρτζεβα, το πρόγραμμα εργασίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2012 με την επιχειρησιακή στρατηγική της Γενικής Διεύθυνσης ΕΚΟ για τον ίδιο χρόνο. Σας υπενθυμίζω ότι αυτό το πρόγραμμα εργασία αποτέλεσε αντικείμενο προηγούμενη συζήτηση με την κυρία Τζόρτζεβα στις 25 Μαΐου και εγκρίθηκε από το ε, Σύνολο των Επιτρόπων 15 Νοεμβρίου του 2012 θα είναι πάρα πολύ σημαντικό έτος στον τομέα τον ανθρωπιστικό δεδομένου ότι προβλέπεται στη μυρίσια διάταξη του προγράμματος η εκπόνηση πρότασης για να μπορέσει να θεσπιστεί ένα ευρωπαϊκό σώμα εθελοντών για την ε, ανθρωπιστική βοήθεια καθώς και η αναθεώρηση της ε, ε, των κανονισμών σχετικά με τα ανθρωπιστικά θέματα που μας είχε προτείνει η Επίτροπος σε μία από τις προηγούμενες δύο. Το 2012 επίσης θα γίνουν και διάφορες συζητήσεις για το επόμενο δημοσιονομικό πολιετές πλαίσιο, με στο οποίο θα πρέπει η ανθρωπιστική βοήθεια να έχει την θέση που τη αξίζει. Αυτή η συνάντηση λοιπόν είναι μέρος επικοδομητικού διαλόγου που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σε συνεχή βάση με ανοιχτό πνεύμα ανταλλαγής απόψεων και ιδεών. Είναι η καταλληλότερη στιγμή για μας για να μπορέσουμε να ανταλλάξουμε ε, ιδέες και γνώσεις για την παρούσα κατάσταση του τρόπου εφαρμογής του προγράμματος εργασίας για την ε, τρέχον έτος και για πολλά άλλα θέματα ε, επίκαιρα σε θέματα ανθρωπιστικά. Σας δίνω μέσα στο λόγο κυρία Επιτροπή. Κυρία Πρόεδρε, ε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, Χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι εδώ σήμερα και χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι σήμερα μάλιστα εδώ που είναι τα γενέθλια της κυρίας Εύα Ζολή και πραγματικά εύχομαι ότι για τα επόμενα 16 χρόνια, για τα επόμενα 60 χρόνια, συγγνώμη, θα είσαστε το ίδιο γεροί και δυνατοί όπως μέχρι τώρα. General overview on where we stand in the... Θα ήθελα να σας δώσω λοιπόν μια γενικότερη έποψη σχετικά με το τι ε, συμβαίνει, ποιες είναι οι αλλαγές οι οποίες θα λάβουν χώρα, καθώς επίσης να σας παρουσιάσω και το πρόγραμμά μας, καθώς επίσης να σας δώσω και μερικά στοιχεία της επιχειρηματικής στρατηγικής ΕΚΟ για την επόμενη χρονιά. πέντε σημεία κλειδιά έχουμε στο επόμενο πρόγραμμά μας, τα οποία θέλα, θα ήθελα σύντομα να σας παρουσιάσω. Η πιο σημαντική προτεραιότητα στρατηγικής ε, και για, και για και για την επόμενη χρονιά είναι βεβαίως η δυνατότητα αντίδρασης ε, στις καταστροφές της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Είχα τη δυνατότητα να σας ενημερώσω για την ε, πρόταση αναθεώρησης του νομικού εργαλείου της προστασίας των πολιτών καθώς επίσης και την ενδυνάμωση της δυνατότητας αντίδρασης σε καταστροφές και την δυνατότητα αναβάθμισης της ε, των δυνατοτήτων που έχουμε όσον αφορά την γρήγορη αντίδραση έτσι ώστε να γίνει ακόμα γρηγορότερο στο μέλλον. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μας στήριξε πάρα πολύ. Η έκθεση Γκαρντίνη ε, που εγκρίθηκε τον Σεπτέμβριο κατά μία έννοια ενισχύει την φιλοσοφία της ε, νομοθετικής μας πρότασης. Αυτό που θέλουμε να επιτύχουμε είναι μεγαλύτερη συνοχή, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, μεγαλύτερη ορατότητα μέσα και έξω σε κάθε είδους καταστροφή. Αυτή τη στιγμή έχουμε ad hoc δέσμευση των κρατών μελών έτσι ώστε από ad hoc να περάσουμε σε εθελοντική μεν αλλά σημαντική δέσμευση αντίδρασης ε, σε καταστροφές έτσι ώστε ανά πάσα στιγμή να ξέρουμε ποια είναι η δυνατότητα επέμβασης που έχουμε. Ελπίζω ότι μέχρι το τέλος ε, τρέχοντος έτους ε, να έχουμε ολοκληρώσει τις διαδικασίες έτσι ώστε να εφαρμοστεί η τροποποίηση και να της νομοθεσίας και να προχωρήσουμε με, με τη διαβούλευση με το Κοινοβούλιο και, την... Ε, και το Συμβούλιο. Δεύτερον, συνένεση για την ανθρωπιστική βοήθεια. Έχουμε προχωρήσει την ενδιάμεση αναθεώρηση, όπως άλλωστε είχαμε προγραμματίσει τον Δεκέμβριο και όπως το είχαμε εγκρίνει το Δεκέμβριο του 2010. Νομίζω ότι κερδίσαμε μέσα από ε, πολλές ε, ε, και επικοδομητικές συζητήσεις και βάσει της έκθεσης Τριφλέρ που έγινε δεκτή από το Κοινοβούλιο τον Ιανουάριο του 2011. Το Συμβούλιο ενέκρινε στα συμπεράσματά του τις τέσσερις προτεραιότητες που είχαμε συστήσει και συνεχίζει η ανθρωπιστική βοήθεια να δίδεται βάσει των ανθρωπιστικών αρχών και των αρχών της ανθρωπιστικής αρρωγής. Επίσης, είναι μεγαλύτερη η αποτελεσματικότητα της ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω ε, εξέβρεσης περισσότερων συνεργειών και βεβαίως συμπεριλαμβάνεται εκεί και η συνεργασία και η ανάπτυξη όταν μιλάμε ε, για ε, καταστάσεις οι οποίες τραβάνε σε μάκρος. Τρίτον, Είμαστε απολύτως δεσμευμένοι με τον Επίτροπο Πίμπελς ε, να αποδείξουμε να αποδείξουμε ότι είμαστε σε θέση, κυρίως σε περίπλοκες καταστάσεις, ε, να αντιδράσουμε. Βεβαίως ε, και στην ακτή του Ελεφαντοστού πρόσφατα έχουμε πάρει σημαντικές αποφάσεις και συμμετείχαμε στις διαδικασίες που εμείς ονομάζουμε «Συνεργασία για τη μετάβαση». έτσι ώστε να μπορέσουμε να επουλώσουμε τις πληγές εκεί που είναι πολύ βαθιές οι πληγές αυτές που έχουν προκαλέσει ε, οι μάχες και τα προβλήματα. Ε, συνεργαζόμαστε βεβαίως με, τις με τα Ηνωμένα Έθνη, αλλά ε, προσπαθούμε να βάλουμε και νέες δωρήτριες χώρες όπως η Τουρκία ή η Βραζιλία στο παιχνίδι. Ε, μας κάνατε μια άμεση ερώτηση πώς είναι δυνατόν ο κανονισμός ε, για την ανθρωπιστική βοήθεια δεν βρίσκεται στο πρόγραμμά μας. Απαντώ. Είδαμε το ενδεχόμενο να αναθεωρηθεί ε, το 2011, ελπίζουμε ότι θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Όμως καταλήξαμε τελικά, όταν ξεκίνησε η διαδικασία, ότι χρειαζόμαστε πρώτα ε, μία πολύ σωστή μελέτη αντικτύπου, καθώς επίσης ε, και την συμπερίληψη όσο γίνεται περισσότερων εμπλεκομένων μερών. Δεν βιαζόμαστε, δεν έχουμε κάποια προθεσμία, ε, δεν εκπνέει οποιαδήποτε προθεσμία δηλαδή θέλουμε να λάβουν χώρα σημαντικές θεσμικές αλλαγές. Έχουμε ήδη την υπηρεσία εξωτερικής δράσης Έχουμε επίσης ε, την ενσωμάτωση της ανθρωπιστικής βοήθειας και της ε, ε, πολιτικής προστασίας και επομένως θέλουμε να είμαστε πολύ προσεκτικοί για το πώς θα αναπτύξουμε τον, το νομικό μας πλαίσιο έτσι ώστε να είναι σωστό και αποτελεσματικό. Και ειλικρινά θέλω να σας πω ότι αισθανθήκαμε ότι υπήρχε επίγουσα κατάσταση όταν φοβηθήκαμε ότι Χάναμε έδαφος όσον αφορά την δυνατότητα παρέμβασης σε μέσω ανθρωπιστικής βοήθειας. Αυτός ο κίνδυνος δεν υπάρχει. Ε, η διαχείριση των ανθρωπιστικών κρίσεων έχει γίνει με αρκετά σωστό τρόπο και επομένως ναι μένει η κατάσταση επίγεια, αλλά παρόλα αυτά δεν αισθανόμαστε να έχουμε ε, κάποια προθεσμία που να μας ε, πιέζει ιδιαίτερα. Γι' αυτό λοιπόν είπαμε ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε με σωστή διαβούλευση, με ανταλλαγή απόψεων, με τις μελέτες που πρέπει να ολοκληρωθούν, έτσι ώστε να ε, προχωρήσουμε σε ένα σύστημα του οποίου η αηφορία και η μακροβιότητα θα ήταν εξασφαλισμένες. Η επόμενη προτεραιότητά μας είναι ε, το εθελοντικό σώμα ανθρωπιστικής ε, παρέμβασης και βοήθειας. Το 2010 είχαμε απομονώσει τα στοιχεία, τα στοιχεία, τα προβλήματα ε, όσον αφορά την ε, χρήση και ανάπτυξη δυνάμεων. Αυτή τη στιγμή έχουμε πιλωτικά προγράμματα έτσι ώστε με πιο σωστό τρόπο να δούμε πώς θα πρέπει να οργανωθεί αυτό το σώμα, αλλά κυρίως ποια δεν θα πρέπει να είναι τα στοιχεία του ε, σώματος αυτού και σε συνεργασία βέβαια και με την εκπόνηση του προγράμματος 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ελπίζουμε ότι μέχρι τα μέσα του επόμενου χρόνου θα έχουμε ολοκληρώσει τις διαδικασίες και πρέπει να σας πω ότι ε, το έτος εθελοντικής εργασίας 2011 μας έδειξε πάρα πολλά ε, ε, νέα στοιχεία σχετικά με το τι ακόμα χρειαζόμαστε όσον αφορά τον εθελοντισμό και την εθελοντική προσφορά. Ε, η συνθήκη για την ε, ε, διατροφική βοήθεια, Food Aid Convention, είναι ένα πολύ σημαντικό επίσης στοιχείο και με μεγάλη χαρά μπορώ να σας πω ότι μετά από έξι διαπραγματευτικούς γύρους που είχαμε φέτους, οι διαπραγματεύσεις έχουν ολοκληρωθεί και ε, έδωσαν και ε, έδωσαν ένα περαιτέρω, μια περαιτέρω όθηση στην επιστημιστική βοήθεια η οποία πέρασε πλέον στον 21ο αιώνα. Νομίζω λοιπόν ότι πλέον μπορούμε να πούμε ότι όσο γίνεται πιο γρήγορα μπορούμε να ενεργοποιήσουμε την συνθήκη αυτή για την επιστημιστική βοήθεια. Επίσης, όπως και για όλους μας και για μας ήταν πάρα πολύ σημαντικό να ε, καταρτήσουμε το, μελλοντικό χρηματοδοτικό πλαίσιο Έχουμε ένα δις ε, ευρώ ανά έτος, εκ των οποίων 915 ε, είναι για την ανθρωπιστική βοήθεια, 30 ε, για το σώμα ανθρωπιστικής βοήθειας και το υπόλοιπο για την προστασία των πολιτών και βεβαίως έχουμε αυξήσει το αποθεματικό από 220 ε, σε 315 εκατομμύρια και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή εμείς ε, ε, προχωρούμε, να μεγαλώνουμε το αποθεματικό αυτό γιατί ξέρουμε ότι οι κρίσεις, οι φυσικές καταστροφές είναι πιο συχνές, είναι πιο σημαντικές, ε, πιο ε, περίπλοκες και επίσης η ανθρωπιστική η ανάγκη ανθρωπιστικής παρέμβασης λόγω ε, των εντάσεων σε ολόκληρο τον κόσμο διαρκώς αυξάνεται και επομένως αυξήσαμε τις δυνατότητές μας έτσι ώστε να ενδύνομαι και τη δυνατότητα παρέμβασης που έχουμε στον τομέα αυτό οι προτάσεις οι οικονομικές που κάναμε έγιναν ε, αποδεκτές ε, πρώτον γιατί ήταν ε, λογικές αλλά και δεύτερον γιατί υπέρ μας μέτρησε το πολύ καλό μητρό που είχαμε και ε, βεβαίω οποιαδήποτε, οποιοδήποτε οικονομικό έλεγχο υπέστημε τον ξεπεράσαμε με, ε, χωρίς να έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε επίσης προσωπικό όχι μόνο στις Βρυξέλλες, πάνω από το 50% του προσωπικού μας βρίσκεται επί τόπου και επομένως ασκούν το καθήκον τους, βρίσκονται εκεί εξ των πολιτών μας να σας πω και δύο λόγια για την επιχειρησιακή στρατηγική μας. Να σας πω λοιπόν ότι τα δύο χρόνια που είμαι επίτροπος, κάτι που έμαθα με τη βοήθεια των συναδέλφων μου είναι ότι εάν χάσουμε μία κρίση, θα γι' αυτό δεν θα μας τιμούνται για τις περιπτώσεις που κάναμε μια σωστή παρέμβαση. Επομένως, η επιχειρησιακή μας αποτελεσματικότητα είναι κάτι που μας απασχολεί πολύ και το παίρνουμε πάρα πολύ σοβαρά. Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε την κάθε κρίση χωριστά, προσπαθούμε μάλιστα ε, να έχουμε όσο γίνεται πιο πρώιμη και πιο γρήγορη ανταπόκριση. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε το, την κρίση στο κέρας της Αφρικής, ε, στο Σαχέλ και γνωρίζετε πολύ καλά ότι το Σουδάν και η Λιβύη ήταν πάντα στις υψηλές μας προτεραιότητες. Και αν δει κανείς τη στρατηγική για το 2012, ε, θα δει ότι καλύπτουμε παρεμβάσεις σε 36 χώρες ή ε, περιοχές μεγάλες ανθρωπιστικές παρεμβάσεις ε, οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι ενεργές και μπορούμε να προβλέψουμε ότι στο, στο Σουδάν ε, στα κατεχόμενα της ε, Παλαιστίνης και στο κέντρο της Αφρικής οι κρίσεις θα συνεχιστούν εάν δεν ενταθούν. Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησής μας θα πάει για μία ακόμα φορά στην Αφρική και στην υποσαχάρη Αφρική 20% για προφανείς λόγους Συνεχίζουμε ε, βεβαίως να ε, οικοδομούμε επί της ε, δημιουργίας υποδομών και δυνατότητας αντίσταση των ίδιων των αντοχή των ίδιων των χωρών και φυσικά 15% των χρημάτων μας θα πάει για μία ακόμα φορά στις παρατηνόμενες κρίσεις, τις παγιωμένες κρίσεις τις οποίες εξακολουθούμε να στηρίζουμε. Θα εντείνουμε την ε, προσπάθεια παρέμβασης που έχουμε όσον αφορά την αποκατάσταση κυρίως ε, σε περιοχές ε, παρατηνόμενης έντασης γιατί θέλουμε να κρατήσουμε ανοιχτές τις προσδοκίες των ανθρώπων και αυτό ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολο αλλά παρόλα αυτά πρέπει να το κάνουμε. Και πρέπει να πω ότι και η πρωτοβουλία της Επιτροπής σας να οργανώσει ε, ειδική ακρόαση για την αποκατάσταση σε αυτές τις περιοχές ε, είναι μια εξαιρετικά καλή πρωτοβουλία. Η επόμενη χρονιά είναι το 20ο γενέθλιο ε, της υπηρεσίας ΕΚΟ, της Εκτελεστικής Επιτροπής και επομένως είναι μια καλή ευκαιρία έτσι ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε πλατφόρμες για να μπορέσουμε με λιγότερα να επιτύχουμε περισσότερα. Καλούμε λοιπόν το Κοινοβούλιο να δράσει μαζί μας έτσι ώστε και να ε, χαιρετήσουμε το γενέθλιο αυτό αλλά και να συνεχίσουμε μαζί τον κοινό αυτό αγώνα. Ευχαριστώ πολύ. Merci beaucoup. Σας πολύ. Το λόγο του κ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήρθα με καθυστέρηση και δεν μπορώ να υποβάλω και αυτό παρά μία ερώτηση που θα συζητήσει με αυτά που πρόλαβα να ακούσω. Αναφερθήκατε στο σώμα των εθελοντών. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν είχατε ανταλλαγή απόψεων με κάποιε οργανώσει με την Κοκόρτ παραδείγματο χάρη, ε, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται το θέμα αυτό. Γιατί κάπω είμαστε ανταγωνιστές θα έλεγα. Και πολλά θα μπορούσαν να συζητηθούν μεταξύ ημών και εκείνων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Στίφλερ. Έχω μια σειρά ερωτήσεων. Εδώθηκαν όμως οι περισσότερες απαντήσει ήδη. Τον περασμένο Νοεμβρίο ήσασταν παρούσα στην πρώτη ανθρωπιστική διάσκεψη στο Παρίσι που οργανώθηκε από τον Γάλλο Υπουργό Εξωτερικών Υποθέσεων που είχε σαν στόχο μια, την οργάνωση μιας ανθρωπιστικής ε, εθνικής βοήθειας σύμφωνα με το ευρωπαϊκό παράδειγμα. Βάσει αυτό που έγινε στο Παρίσι, πιστεύετε ότι κάτι τέτοιο θα μπορεί να οργανωθεί και θα μπορούσε η Κομισιόν να αναλάβει την πρωτοβουλία για να μπορέσει να γίνει καλύτερη γνωστή όσον αφορά τη συνένεση. Μου φαίνεται ότι εκεί υπάρχει κάποιο κενό από πολλά κράτη-μέλη. Και κατόπιν έχω μια ερώτηση όσον αφορά την ησυχία που έχουμε όλοι για τη Συρία αυτή τη στιγμή. Αλλά νομίζω ότι απαντήσατε. Και για να δω, για να δω, να συγχωρείτε. Ναι, ναι. Όσον αφορά την Κένια, όπου πρόσφατα είχα πάει. Η Γενική Διεύθυνση εγώ, ε, επειδή πολλά στις ε, ε, ξηρές και ημιξηρές περιοχές της χώρας. Δεν ξέρω κατά πόσον αυτό είναι θέμα ανάπτυξης ή υπάρχει και ένα συμφέρον τη κυβέρνηση και των εταίρων εκεί τη ανάπτυξη αυτών των περιοχών και έλλειψη οργανωμένης αντιμετώπισης της ε, λειψιδρίας. Είναι θέμα κρίσης ε, επίγουσας, είναι θέμα μακροπρόθεσμης κρίσης και πώς πιστεύετε ότι η ανθρωπιστική βοήθεια και η αναψιακή βοήθεια μπορούν να συνδυστούν. Γιατί ξέρετε ότι εσείς είχατε πάει πριν από μήνε μήνες σε αυτή τη χώρα, στην Κένια. Ευχαριστώ κυρία Κέλλα, έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Εγώ θα ρωτήσω κάτι όσον αφορά το συσχετισμό μεταξύ ε, της ενίσχυσης για ανθρωπιστική και ανθρωπιστικούς λόγους και της αναπτυξιακής βοήθειας. Εσείς πώς πιστεύετε ότι αυτός ο συσχετισμός μπορεί πραγματικά να διαφανεί ξεκάθαρα στα δημοσιονομικά μέσα. Και το δεύτερο ερώτημα αφορά τις κλιματικές αλλαγές που βέβαια όσο πάει επιδεινώνεται πολλού από, τους, ε, από τις καταστροφές με τις οποίες έχετε να κάνετε εκεί. Λαμβάνετε υπόψη στις προτάσεις που θα υποβάλλετε του χρόνου το θέμα αυτών των κλιματικών αλλαγών. Και τέλος, ε, ε, σε αυτό που είπατε για την πρόληψη, όπως είδαμε, πολλές από αυτές τις κρίσεις μπορούν πραγματικά να μειωθούν, όχι να αποφευχθούν. Βέβαια, να να αποφευχθούν με κάποια πρόληψη. Εκεί ίσως κάτι μπορούσατε να μου πείτε πραγματικά. Ευχαριστώ. Κυρία Γεωργίευα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κάνουμε κάτι καλύτερο από το να, μην μιλάμε, από το να μιλάμε στους εκπροσώπους των μη κυβερνητικών μας ε, οργανώσεων τους. Είπαμε να συμμετάσχουν στον όλο σχεδιασμό των ε, δράσεων μας. Υπάρχουν πιλωτικά προγράμματα με την Ερυθρό Σταυρό, με το Save Children στο Ηνωμένο Βασίλειο, με θελοντικές οργανώσεις, διότι αυτό που δεν θέλουμε να κάνουμε είναι να δαπανίσουμε χρήματα για κάτι το οποίο ήδη έχει αναλυφθεί από άλλους. Θέλουμε να κάνουμε κάτι εκεί που πραγματικά είναι αναγκαίο, απαραίτητο να γίνει και έχουμε εντοπίσει ότι υπάρχουν δύο μεγάλες αδυναμίες, δύο κενά. Πρώτα απ' όλα, ετοιμότητα και πρόληψη. Υπάρχουν όσον αφορά την αντίδραση πολλές μη κυβερνητικέ γνώσεις. λίγες όμως έχουν τις δυνατότητες, τις δεξιότητες και την ικανότητα να αποδείξουν ότι έχουν προληπτική δύναμη λαμβάνοντας μέτρα όπως φερειπίν η αναδάσταση αναδάσωση, ε, διαχείριση υδάτινων πόρων και πολύ αλλά σε κοινοτικό επίπεδο. Και τώρα θα επανέλθω σε αυτό να μιλήσω για τις κλιματικές αλλαγές. Δεύτερο πρόβλημα που υπάρχει και το πείσαμε. Δυνατότητα διαχείρισης των ε, ειδικοτήτων ε, ταχείας και επίγουσας αντίδρασης. Όλοι σχεδόν παραπονούνται ότι όταν υπάρχει μια πολύ σημαντική επίγουσα κατάσταση, πάρα πολύ λίγα άτομα επιτόπου είναι αυτά τα οποία μπορούν να προσφέρουν σε τέτοιου είδους ε, καταστάσεις ε, τις γενικές κατευθύνσεις πρέπει να ακολουθηθούν, που μπορούν να διαχειριστούν τέτοιου είδους καταστάσεις. Η κατάρτιση, διότι έχουμε την εντύπωση ότι πιο τυποποιημένη και απλή και κατανοητή κατάρτιση είναι απαραίτητη. Αύξηση του ποσοστού θελοντών ε, σε χώρες στις οποίες υπάρξει, υπάρχει έλλειψη, διότι εμείς στην Ευρώπη, όσον αφορά τον εθελοντισμό, το πάμε πολύ καλά. 400.000 εθελοντές ετησίως έχουμε. Αυτός πρέπει να πω ότι δεν είναι ε, μια δραστηριότητα την οποία επιμερίζονται κατά ίσο τρόπο οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Παίρνουν χώρες τις οποίες έχουμε 40% ποσοστό, ε, σε άλλες λιγότερο από 10. Στη χώρα μου φανταστείτε 6% είναι το ποσοστό Και φανταστείτε στην παλιά εποχή του κομμουνισμού ε, ήταν υποχρεωτικό να είναι σε εθελοντή. έτσι δημιουργήθηκε μια επιδερμική και αλλεργική αντίδραση, αν θέλετε, προ τον ε, εθελοντισμό. Εγώ για πρώτη φορά ήμουν εθελόντρια, κύριε Πρόεδρε. Υποχρεώθηκα να είμαι εθελόντρια για πρώτη φορά όταν ήμουνα ε, στα πρώτα χρόνια του Πανεπιστημίου. Λυπάμαι, θυμάμαι λοιπόν ε, τρομερά πράγματα. Πραγματικοί σκλάβοι είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε κάτι. Και ήμουνα σε ένα εργοστάσιο επεξεργασία ειδών διατροφής ε, σε ένα εργοστάσιο και ποτέ πρέπει να πω στη ζωή μου δεν θα δοκιμάσω τα τρόφιμα που παρήγαγε αυτή η βιομηχανία. Και για να μπορέσω να ξεφύγω έγινα αθλήτρια. Καταλαβαίνετε λοιπόν πώς είναι το θέμα. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ε, μία προσδοκία, μία φιλοδοξία με τον ατόμων που θέλουμε να προσελκύσουμε, ότι αυτό που θα κάνουν θα είναι κάτι καλό για να μπορέσουμε να παράσχουμε τέτοιου είδους υπηρεσία. Επίσης, θα ήθελα να πω το εξή στην κυρία Στίφλερ. Πρώτα απ' όλα πάρα πολύ ειλικρινά να εκφράσω και την ευγνωμοσύνη μου στην Γαλλία και στον Υπουργό κ. Ζιπέ που οργάνωσε αυτή τη διάσκεψη, διότι ήταν ένα μήνυμα ότι ακόμη και σε αυτή την δύσκολη οικονομική περίοδο για την Ευρώπη, εμείς εδώ βρίσκουμε και χρόνο για να συζητήσουμε για αρχές και για αξίες. Ποιος ήταν ο στόχος αυτής της διάσκεψης, να επαναλάβει την ε, δέσμευση της Γαλλίας για την προσέγγιση της Γαλλίας όσον αφορά την ανθρωπινική βοήθεια. Και η σύσταση ότι πρέπει να κάνουμε κάτι στα 20 χρόνια της ΕΚΟ είναι πολύ σωστή. Κάτι θα οργανώσουμε ώστε να μπορέσουμε να ευαισθητοποιήσουμε περισσότερο ε, τον κόσμο όσον αφορά τις ε, αρχές της ανθρωπιστικής βοήθειας που θα πρέπει να μας διαπρόσουν, όσον αφορά την γένεια. Σωστά τα είπατε στην ΕΚΟ ε, η πιλωτική μελέτη έδειξε ότι οι δραστηριότητες που μειώνουν τον κίνδυνο είναι πρωταρχική σημασία. Το ποσοστό ε, κακής διατροφής μεταξύ των παιδιών στην περιοχή αυτή της Κέννης ήταν 50% χαμηλότερο από ό,τι στις άλλες περιοχές δεδομένου ότι από το 2006 είχαν γίνει διάφορες δραστηριότητες για να μπορέσουν να είναι πιο ανθεκτικοί οι άνθρωποι και κυρίως να προσθέτουν τα παιδιά σε περίοδο τρομερής ξηρασίας. Ο Επίτροπος Πίμπαλς έλαβε μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία για την ε, αντίσταση στην ε, περιοχή του κέρατος της Αφρικής και πιστεύουμε ότι υποστηρίζουμε τις δραστηριότητες και θέλουμε θα πρέπει αυτά τα προγράμματα αντίσταση τέτοιου είδους ακραίες καταστάσεις να μπορέσουμε να τα εφαρμόσουμε σε αυτή την περιοχή και σε άλλες περιοχές που είναι ευάλωτες σε θέματα φυσικών καταστροφών. Και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει άμεση σχέση με το να συνδέσουμε την πολιτική μέτρων ανακούφισης με την πολιτική που ακολουθούμε για να βοηθήσουμε τις χώρες αυτές. Κυρία Κέλλερ. Στα πλαίσια των ε, πολιετών δημοσιονομικών ε, προσαρμογών προβλέψεων Είμαστε αποφασισμένοι ότι ε, κάνουμε να το κάνουμε με τρόπο που να είναι ορατός στους άλλους, να φαίνεται ακριβώ κάνουμε. Πώς? Ή θα θεσπίσουμε στόχους που τον οποίο η υλοποίηση μπορεί να εποπτεύεται από κάποιον, διότι θα πρέπει να είμαστε υπόλογοι και να φαίνεται αυτό. Εγώ θα προτιμούσα να έχουμε ένα δημοσιονομικό μέσον για το σκέλος ανάπτυξη που να είναι πιο ευέλικτο και να μπορεί να αντιμετωπίζει τις ανάγκες και τους στόχους ανάπτυξης συνεχώς, σε συνεχή βάση. Για να εξηγηθώ. Ε, ό,τι αφορά το ανθρωπιστικό σκέλος μπορεί να γίνει αρκετά γρήγορα δεδομένου ότι εμείς δεν δίνουμε χρήματα σε καμία κυβέρνηση, το δίνουμε σε εταίρους, σε συνεργάτες που έχουν αποδείξει ότι έχουν την δυνατότητα να ανταποκριθούν σε ένα συγκεκριμένο μέρος σε αυτό το οποίο ζητείτε. Αλλά όταν τελειώσουμε το ανθρωπιστικό σκέλος και σώσουμε τις ανθρώπινες ζωές, κατά κάποιο τρόπο αποτραβιόμαστε και δεν παρακολουθούμε του σύνεγγες τι γίνεται για την ανάπτυξη περαιτέρω Θα ήθελα λοιπόν εγώ να έχουμε ένα δημοσιονομικό μέσο που θα επιτρέπει πέραν του τι κάνουμε εμείς το ανθρωπιστικό σκέλος, σύντομα να μπορεί να προσδίδει και κάποιους οικονομικούς πόρους που βοηθήσουν την ανάπτυξη. Γι' αυτό στην καλύτερη των περιπτώσεων λέμε ότι ας δούμε ποια είναι τα καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα που μπορούμε να επιτύχουμε όταν ολοκληρώσουμε την πρώτη φάση του έργου μας. Και τώρα, όσον αφορά τις κλιματικές αλλαγές, η αντιμετώπιση των προβλήματος είναι παρεμφερής, θα έλεγα. Τι κάνουμε. Η δουλειά που κάνουμε θέλουμε να εμπνεύσει και άλλους. Διότι είδαμε πόσο καταστροφικά μπορεί να αποτελέσουν το κλιματικών αλλαγών. Διότι η φυσικές καταστροφές είναι καταστροφές που ε, μπορεί ο καθένα να αντιμετωπίσει. Η δική μας λοιπόν ευθύνη είναι να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις κλιματικές αλλαγές και να κάνουμε τον κόσμο πιο ανθεκτικό. Και μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Στην Ευρώπη, σε κάθε επόμενο κανονισμό θέλουμε ό,τι κάνουμε να μπορεί να ανθίσταται κατά κάποιο τρόπο στις μεγάλες αυτές ειδικές καταστροφές. Το ίδιο και όσον αφορά την πολιτική μας για την ε, ανάπτυξη και τη συνεργασία. Δυστυχώς η επιτυχία όμως εξαρτάται από το αν υπάρχει συμφωνία μεταξύ όλων. Πράγμα το οποίο δεν είναι εύκολο να υλοποιηθεί. Μπορώ να πω για την Ευρώπη ότι η Ευρώπη δεν θα πρέπει να υιοθετήσει την εξή στάση. Η αδυναμία των άλλων είναι για μας πρόσχημα να μην κάνουμε κάτι σωστά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Τώρα. Ο κύριος Νόισερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε. Σας άκουσα με ενδιαφέρον, γιατί έχουμε ρίξει ότι αυτά που μας είπατε σήμερα είναι κάπως και στο πρόθεσμο απολογισμός της εργασίας μας και είναι ένας απολογισμός ο οποίος πραγματικά είναι πολύ αξιόλογος μετά από δύο χρόνια. Με πείθη Είναι πολύ πιστική η εργασία σας και έχει όλες τις προοπτικές για το μέλλον μέσα της. Χαίρομαι που στην αντιμετώπιση της κρίσης λαμβάνεται υπόψη δύο πράγματα. Την πρόληψη των κρίσεων αφενός και την ε, συνοχή που δίνεται, όπως το παράδειγμα για την δεχτή του ελεφαντοστού. Υποθέτω και στο κέρας της Αφρικής ε, η κατάσταση θα ήταν παρόνια. Τα πα, παραδείγματα τα ίδια και ως μέλος ε, αντιπροσπέζει για την Παλαιστίνη χαίρομαι που αναφερθήκατε και στην Παλαιστίνη. Πολιετή προγραμματισμό, αυτή η κατανομή σε ανθρωπιστική βοήθεια ε, βοήθεια για φυσικές καταστροφές και ε, χρηματοδότηση μακροπρόθεσμα είναι σωστή. Αλλά πώς θα γίνει η ιεραρχία είναι κάτι που θα πρέπει να το δούμε ίσως εκ τον υστέρων. Και είναι πολύ καλό που υπάρχει και ένα αποθεματικό το οποίο όσο πάει και αυξάνεται και δίνει τη δυνατότητα πόρους που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί το ένα έτος ε, να μεταφέρονται στο επόμενο. Έτσι η βοήθεια είναι πολύ πιο αποτελεσματική. Και αυτό το έχει εκτιμήσει και θετικά και το ηλεκτρικό συνέδριο στα πλήρε της εργασίας σας. Η ερωτήση μας είναι εξής. Αναφέρατε ότι χρειάζεται πολύ συντονισμός. Πρέπει να είναι τεράστιο το έργο αυτό. Αλλά ότι θέλετε να συντονίσετε ακόμα περισσότερο τη συνεργασία και με τους άλλους ε, χρηματοδότες, αραβικές χώρες, Βραζιλία, Κίνα, είναι πάρα πολύ σημαντικό νομίζω, γιατί εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούμε ότι είμαστε στο επίκεντρο της ε, ε, βοήθειας ε, σε περιπτώσει καταστροφών με τη σύπα ίσως μαζί. Λοιπόν, ποια θα είναι η μορφή του συντονισμού αυτού στο μέλλον. Και επίσης, η Επιτροπή μας νομίζετε ότι μπορεί να σας στηρίξει. Εγώ πολλέ φορέ αισθάνομαι ότι είμαστε ένα μονομάχο, ότι είμαστε ένας μονομάχος εδώ και είναι καλό να μπορέσουμε να συνεργαστούμε και εάν μα χρειαζόσετε πέστε μα πού μπορούμε να σα βοηθήσουμε για να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα από κοινού. Ευχαριστώ. Ο κύριο Τζούτουντάν, παρακαλώ. Μάλιστα, πρόεδρε. καμία απογοήτευση, την αναφέρατε όμως. Είναι το θέμα της αναθεώρησης των περιεσιών ανθρωπιστικής βοήθειας. Τα σχόλια σας μου έδωσαν την εντύπωση ότι υπάρχει μια πλήρης μελέτη αντικτύπων. Δηλαδή τι, αναβλήθηκε ΣΑΗ ή θα γίνει α, του χρόνου ή τουλάχιστον όσο είστε στις Επίτροπος ή πότε θα γίνουν όλα αυτά. Ευχαριστώ κυρία Ντεκάιτσερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, εν μέρει απαντήσατε στις ερωτήσεις που είχα όσον αφορά το σχετισμό ε, μεταξύ της ε, ε πήγουσας βοήθειας και άλλου τύπου βοήθειας σε ορισμένε χώρες γιατί σε περιπτώσεις όπως η Κένια, η Σομαλία, ιδίω και άλλες χώρες βλέπουμε ότι υπάρχει πραγματικά ένα συσχετισμός μεταξύ των δύο και κανένα ασχολείται μόνο με μια μικρή πτυχή όταν εξετάει μόνο το κατεπήγον, αλλά εξετάσε το θέμα της διακυβέρνησης των μοντέλων ανάπτυξης που επιβλήθηκαν στις χώρες αυτές που δεν είναι σίγουρα ανάλογες με τις τοπικές ανάγκες. Όλα αυτά είναι ένα σύνολο. Εγώ θα ήθελα να σας υποβάλω μια ερώτηση πάνω στο εξή. Ποια είναι η λύση που βρίσκετε εσείς ε, σχετικά με τις δυσκολίες πρόσβασης στην ε, επίγουσα βοήθεια. Παραδείγματο η βοήθεια που δίνεται σε ορισμένες περιοχές ε, μετά από βομβαρδισμούς είναι πολύ δύσκολο οι πληθυσμοί εκεί να έχουν πρόσβαση στη βοήθεια αυτή μετά από βομβαρδισμούς. Στη Σομαλία το ίδιο, τι γίνεται κάτω από πολύ δύσκολες πολιτικές αυτό το Θέμα δηλαδή της πρόσβασης σε αυτή τη βοήθεια που είναι πάρα πολύ σημαντική. Πώς το βλέπετε. Και όσον αφορά την ε, δημοκρατική δημοκρατία του Κονγκό, προβλέπετε κάτι. Γιατί και εκεί επίκυνε κάποιες ανθρωπιστικές καταστροφές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Γεωργίευα, έχετε το λόγο για να απαντήσετε στις ερωτήσεις αυτές. Ευχαριστώ πολύ. Προφανώς δεν ξεχνώ ότι η θητεία μου είναι πενταετής. Κατά κάποιο τρόπο βρισκόμαστε πλέον στα μισά του δρόμου. Έχουν περάσει ήδη δύο χρόνια. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει κανείς να έχει πολύ σαφείς στόχους σχετικά με το τι θέλει να πετύχει το επόμενο μισό. Για το θέμα αυτό που θίξατε υπάρχει και προβλέπεται και ειδική συνάντηση. Βεβαίως μου λένε ότι τα τελευταία, το τελευταίο καιρό δεν ε, μπορούν να αναλυφθούν ε, νέες ε, πρωτοβουλίες, αλλά δεν είμαστε ακόμα στον τελευταίο καιρό, έχουμε ακόμα δύο χρόνια μπροστά μας. Και προτιθέμεθα να υπογραμμίσουμε περισσότερο το ε, κομμάτι της πρόληψης, της ανάπτυξης ε, της ανθρωπιστικής βοήθειας ε, και της ανακούφισης που αυτή μπορεί να προσφέρει. Βεβαίως να αυξήσουμε και τον αριθμό των δωρητών έτσι ώστε τα ποσά να αυξηθούν. Βεβαίω τα Ηνωμένα Έθνη θα πρέπει να μπουν στο παιχνίδι, αλλά εξ ορισμού οτιδήποτε ε, ε, κάνουμε για να ενδυναμώσουμε την θέση των Ηνωμένων Εθνών ε, ταυτόχρονα αυξάνει το ποσοστό των δωρητών. Συζητούμε και με τη Ρωσία και με την Κίνα, με την Τουρκία, σας το είπα και προηγουμένως, και επίσης και με τον Αραβικό Σύνδεσμο, έτσι ώστε να βρούμε νέους δωρητές. Ένας είναι ο στόχος μας να διασφαλίσουμε ότι όλοι κατανοούμε το ίδιο πράγμα. Δηλαδή ότι η ανθρωπιστική βοήθεια δεν είναι πολιτική. Δηλαδή ότι δεν έχει κανείς διαφορετικούς τρόπους για να ε, ε, αντιμετωπίσει ανθρωπιστικές ε, κρίσεις. Βοηθάμε τους ανθρώπους εκεί που έχουν ανάγκη τη βοήθεια. και προσπαθούμε να επιτύχουμε αυτή τη σταθερότητα η οποία μόνο καλά αποτελέσματα μπορεί να φέρει σε κάθε επίπεδο και να βοηθήσει τον κόσμο. Πιστεύω ότι μέχρι τώρα το Κοινοβούλιο υπήρξε εξαιρετικά ε, καλός βοηθός μας ας πούμε όσον αφορά την ε, ικανότητα αντίδρασης ε, σε ε, φυσικές καταστροφές στην, στον τομέα της διασύνδεσης, της προστασίας με την αποκατάσταση, της αντιμετώπισης της κρίσης δηλαδή με την αποκατάσταση. Έχουμε πάντα αργό το κοινοβούλιο και αυτό πραγματικά είναι μεγάλη δύναμη για την ομάδα μας. Τώρα, εάν υπάρχουν ειδικά εξειδικευμένα προβλήματα, βεβαίως θα στραφούμε πάλι σε εσά για να μας βοηθήσετε. Όσον αφορά το ερώτημα, το εάν θα τελειώσουν αυτά στη δικιά μου θητεία, ναι, ναι, σίγουρα. η αξιολόγηση που κάναμε ήταν εξαιρετικά προσεκτική. Και όταν αποφασίζουμε ότι κάτι το φάζουμε στις προοπτικές μας, σημαίνει ότι το έχουμε μελετήσει πολύ προσεκτικά. Και βεβαίως ε, η ακεραιότητα και η αμεροληψία της ανθρωπιστικής βοήθειας είναι εκ των ουκάνευ. Και θέλουμε να προωθήσουμε ακόμα περισσότερο τη συζήτηση αυτή. Τώρα που πλέον ε, δεν ε, διαφαίνεται ο κίνδυνος αυτός και που ε, το, το επίγον του πράγματος έχει περάσει, νομίζω ότι είναι πιο σόφρονο από την πλευρά μας να σκεφτούμε περισσότερο. Να δούμε, να συζητήσουμε όλες οι πλευρές και αυτό βεβαίως παίρνει περισσότερο χρόνο. Πάντως, σας υπόσχομαι ότι δεν πρόκειται να φύγω από τη θέση αυτή εάν δεν ολοκληρώσω τη διαδικασία αυτή. Και βεβαίως μπορεί να προχωρήσω και σε μια δεύτερη εντολή, άρα κανένα πρόβλημα. Όσον αφορά το θέμα των φόρων. Για την ανθρωπιστική βοήθεια υπάρχουν μονάχα δύο προϋποθέσεις, δύο όροι. Ένα, Πρώτος όρος, να είναι ε, σαφής η ανάγκη και δεύτερον να μπορούμε να φτάσουμε ε, στους ε, στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. αυτή είναι οι άξονες πρόσβασης που έχουμε. Και προχωρούμε με τρεις τρόπους. Πρώτον, δουλεύουμε με εταίρους οι οποίοι έχουν αποδείξει ότι επιτυχημένα μπορούν να ε, δραστηριοποιηθούν σε ένα εξαιρετικά σταθές περιβάλλον. Ο κόσμος είναι ε, μικρός όσον αφορά αυτό το θέμα. Το ICRC συνεργαζόμαστε με το ICRC ή μάλλον όχι, να τα πω καθαρίτερα στη, ο έλεγχος όχι της Σομαλίας ολόκληρης, αλλά της περιοχής Al-Shabaab. Η περιοχή Al-Shabaab, από την οποία εκδιώχθησαν πρόσφατα 16 μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι ότι η πρόσβασή μας έχει μειωθεί τη στιγμή που οι ανάγκες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Access. And as στο Μπουνάου είναι, είναι σχεδόν ε, αδύνατη η πρόσβαση. Εμείς δεν θέλουμε αυτήν την λεγόμενη ε, ε, διασυνοριακή συνεργασία. Δεν θέλουμε να δώσουμε τα χρήματα των φορολογούμενων χωρίς να ξέρουμε, χωρίς να ξέρουμε πού πάνε και πώς θα χρησιμοποιηθούν. Επομένως, σε μερικές περιπτώσεις είναι γεγονός ότι είναι μηδαμινή η δυνατότητα βοήθειας που έχουμε. Επομένως, θέλουμε οργανώσεις οι οποίες να έχουν βρει τρόπο να φτάσουν μέχρι τον ε, κόσμο. Θέλουμε συνεργασία με κυβερνήσεις έτσι ώστε να έχουμε διασφαλισμένη πρόσβαση. Και τρίτον, βοηθούμε αυτούς που καταφέρνουν να ε, εγκαταλείψουν τις περιοχές ως πρόσφυγες. Δεν είναι όλα καλά βέβαια. Αλλά μας θυμίζει κιόλας το γιατί δεν θέλουμε να έχουμε αποτυχημένες, ε, αποτυχημένα κράτη ή αποτυχημένες περιπτώσεις όπως τη Σομαλία ας πούμε που είναι μια χαμένη περίπτωση. Η ανθρωπιστική αντίδραση δεν αποτελεί λύση του προβλήματος γιατί το θεμελιώδες πρόβλημα είναι εκεί, στο αποτυχημένο κράτος και ε, ε, ε, εδώ βεβαίως σε αυτές τις περιπτώσεις χρειαζόμαστε, στα αποτυχημένα κράτη, χρειαζόμαστε πιο ολοκληρωμένη παρέμβαση. Η κυρία Δεκεζέρ. Κύριε Επίτροπε, μία παρατήρηση. Ασκήσατε πια στην κυβέρνηση για να έχετε πρόσβαση πάρα πολύ δύσκολες περιπτώσεις. Στην περιοχή του Blue Nile, στην περιοχή της είναι καταστροφική η κατάσταση. Είδα τον νέο πρέσβη του Σουδάν στο Χαρτούμ, ο οποίος μου μίλησε γι' αυτό το σχέδιο ανάπτυξης της ανατολικής πλευράς κτλ. και, Και λέει ότι θα προχωρήσει αυτή το σχέδιο ε, αφήνοντας κατά μέρος την περιοχή Blue Nile και Blue Mountain. Πώς είναι δυνατόν να γίνει έτσι, να προωθήσουμε προς αυτή την περιοχή αναπτυξιακή βοήθεια, ενώ δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για την περιοχή Blue Nile. Δεν καταλαβαίνω. Εκεί δεν έχουμε πρόσβαση. Τι μπορούμε να κάνουμε. Θα ήθελα και εγώ, λέει η Πρόεδρος, να κάνω δύο ερωτήσεις η Ευρώπη παρεμβαίνει σε όλα τα μετανασταυτικά ρεύματα και τα ε, ε, στρατόπεδα συγκέντρωσης τα οποία υπάρχουν άτομα μετά την ε, Αραβική Άνοιξη. Στην περίπτωση της Συρίας ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποια στρατόπεδα προσφύγων και στην Τουρκία μετά τα γεγονότα της Συρίας. Τι ανάγκες υπάρχουν εκεί. Εγώ πριν από μερικές μέρες επισκέφθηκα το πολύ απομακρυσμένο διαμέρισμα της Γαλλίας, τη Μαγιότ. Δίπλα στις Κομόρες. Συζήτησα με διάφορες μη κυβερνητικέ οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μου είπαν ότι υπάρχουν ετησίως εκατοντάδες άτομα τα οποία βρίσκονται στη θάλασσα μεταξύ Μαγιότ και Κομόρ. Μπορούμε να κάνουμε κάτι, υπάρχει κάποιο πρόβλημα για να μπορέσουμε όσοι σώζονται και είναι πρόσφυγες σε αυτή την περιοχή να βοηθηθούν. Και η κυρία Κέλλαρ και πάλι ζήτησε το λόγο. Για να συνεχίζω σύντομα ε, αυτό το οποίο ελέγχθηκε για την συνεργασία ε, μεταξύ Επιτροπής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όν; θα ήθελα να αναφέρω ότι θα θέλατε να υπάρχουν πιο ευέλικτα μέσα στα δημοσιονομικά μέσα για να μπορέσει να υπάρχει ταχύτερη ανταπόκριση σε περίπτωση καταστροφής και ανάπτυξης μεταξύ αυτών των δύο. Μπορείτε, μπορείτε να μας πείτε με περισσότερη ακρίβεια τι προβλέπετε, τι θα γίνει. Αυτό το μέσον θα είναι μέλος του DCI, θα είναι κάτι το διαφορετικό τα ποσά που θα χρησιμοποιηθούν θα μπουν στο αποθεματικό, πώς προβλέπετε να διαμορφωθεί αυτή η πολιτική που θέλετε. Όσον αφορά το Blue Nile, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι στην πλευρά ανθρωπιστικής βοήθειας είμαστε υποχρεωμένοι να βοηθούμε τα άτομα εξαιτίας των αναγκών που έχουν. Δεν επιβάλλουμε κυρώσεις στα άτομα, διότι υπάρχουν ε, αδυναμίες και προβλήματα στις κυβερνήσεις. Παρέχουμε βοήθεια, φαρμακευτική, προστασία, ε, στέγαση στα άτομα τα οποία έχουν επηρεαστεί άμεσα από αυτού του είδους την πολιτική. Στο Σουδάν, στο Χαρτούμ, στη Τζούμπα. Πολύ άσχημα πράγματα συμβαίνουν και όλο και περισσότερο υποφέρουν. Τι προσπαθούμε να κάνουμε, να φτάσουμε σε αυτά τα άτομα πρώτα απ' όλα και αυτοί που παρέχουν τη βοήθεια πολλές φορές δεν έχουν πρόσβαση. Ποια είναι η λακτική λύση. Να στέλνουμε διασυνοριακά χρήματα. Και δεν ξέρουμε πού πηγαίνει αυτή η βοήθεια. Δεν ξέρουμε σε ποιον φτάνει, αλλά την αποστέλουμε ούτως ή άλλως. Στις συζητήσεις που κάνουμε υπάρχουν πάρα πολλές επιφυλάξεις όσον αφορά αυτή την προσέγγιση, όπου δεν υπάρχει υπόλογος και υπεύθυνο από την άλλη μεριά. Και ξέρουμε, δεν ξέρουμε τι γίνονται τα χρήματα, μήπως σκοτώνονται περισσότεροι, μήπως γίνονται περισσότερο αρνητικά πράγματα, δεν ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Όταν λοιπόν ανέφερα την πρόσβαση Γι' αυτό είπα ότι είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Διότι μπορώ να σας πω, ακούστε, αυτό ε, κάνουμε για να βοηθήσουμε, να βοηθήσουμε τα διάφορα άτομα που υποφέρουν. Αλλά σήμερα πάρα πολύ λίγα μέρη στον κόσμο έχουν τόσο δύσκολη η αδύνατη πρόσβαση όπως η περιοχή του Blue Nile. Μέρος της Ομαλίας, Νότιο Σουδάν. Και εάν η αποχωρήσουν, ή, συγγνώμη, αν συμμετέχουν και άλλες οργανώσεις του ΟΗΕ και εμείς εκεί είμαστε. Όπως ο Ερυθρός Σταυρός, με τον οποίο έχουμε με τη Διεθνή Επιτροπή του Σταυρού πάρα πολύ καλή συνεργασία. Αλλά, επαναλαμβάνω, δεν έχουμε πλήρη πρόσβαση. Τώρα, όσον αφορά το TRC. Έχουμε 44 εκατομμύρια ευρώ για ανθρωπιστική βοήθεια, ενώ οι προβλεπόμενες ανάγκες, ξέρουμε ποιες είναι, ξέρουμε ποιοι είναι οι εταίροι που πρέπει να μας βοηθήσουν. Αλλά έχουμε θέση εκκίνηση και έναν μηχανισμό ε, προστασίας ανθρωπιστικής εκ των προτέρων, ώστε να είμαι σε ετοιμότητα και αν χρειαστεί να μπορέσουμε να εκενώσουμε κάποιες περιοχές, να μπορέσουμε να το κάνουμε ανάλογα με το πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Και βεβαίως παρακολουθούμε και τις εξελίξεις για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε έγκαιρα. Όσον αφορά τη Συρία, προφανώς το πρόβλημα στη Συρία έχει ξεπεράσει τις ε, καταχρήσεις σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχει μία μεγάλη διάσταση ανθρωπιστική, διότι ξέρουμε ότι πολλά άτομα προσπαθούν να εγκαταλείψουν τη Συρία, αλλά και εντός της Συρίας έχουμε άτομα στην Δαμασκό εξαιτία των προσφύγων από γειτονικέ χώρες. Αλλά αυτό που μπορώ να πω ότι είναι ο τρόπο το οποίο μπορούμε να ενεργήσουμε πολύ περιορισμένο. Όσον αφορά την Τουρκία. Σχεδιάζω να επισκεφθώ την Τουρκία σε αρχές ε, του επόμενου έτους και θα επισκεφθώ του τα, τους καταβλισμούς των προσφύγων και θα δω επιτόπου περί τίνος πρόκειται. Βεβαίω, τα πάντα εξαρτώνται από τι αρχέ τη Τουρκία, αν θα μπορέσουν να οργανώσουν μία και θα επιτρέψουν μια τέτοια επισκέψη. Αλλά αρχέ του επόμενου θα το κάνω αυτό το ταξίδι. Τώρα, σαν αφορά το πρόβλημα των μεταναστών. Αυτό είναι θέμα αρμοδιότητας Επιτρόπου Μάλστρομ. Όταν έχουμε μετανάστευση εντός της Ευρώπης, είναι υπεύθυνη η Επίτροπος Μάλστρομ. Και παρέχεται στα κράτη-μέλη μια κάποια βοήθεια όταν αντιμετωπίζουν ε, μεγάλες εισρωές μεταναστών. Και πρέπει να πω ότι όντως πρόκειται για ένα σοβαρό πρόβλημα. Αλλά πολλές φορές βλέπουμε μόνο την αιχμή του δώρατος, δεδομένου ότι πάρα πολλά άτομα τα οποία μετακινούνται εσωτερικά, είναι πρόσφυγες, βρίσκονται στις ε, ε, αναπτυσσόμενες χώρες. Πέρσι η Νορβηγική η Αρχή που με αυτά τα θέματα μας ανέφερε ότι υπάρχουν 240.000 μετακινούμενες στο Ρεκάνδα και 90% των κινήσεων αφορούν κινήσεις ανθρώπων από μία πολύ λίγο αναπτυγμένη χώρα από μια άλλη. Πρέπει να δούμε λοιπόν πώς θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Και βεβαίως η κλιματική αλλαγή προσθέτει και επιβαρύνει αυτό το πρόβλημα, διότι οι πρόσφυγες λόγω κλιματικών αλλαγών είναι πλέον μια νέα ειδική κατηγορία. Η Νορβηγία οργάνωσε μια πολύ ε, μεγάλη συνάντηση όπου συζητήθηκαν αυτά τα προβλήματα. Διότι πρέπει να δούμε πώς θα προσεγγίσουμε αυτό το θέμα των μακροχρόνια προσφύγων που είναι δικό μας θέμα, δική μας αρμοδιότητα όταν απειλούνται οι ζωές τους και πρόκειται για ανθρωπιστικό πρόγραμμα. Πρόβλημα. Και βεβαίω εδώ αναφέρομαι για του πρόσφυγε οι οποίοι βρίσκονται σε αναπτυσσόμενε χώρε και όχι αυτού που μπαίνουν στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ε, ανταλλαγή απόψεων. Θέλετε να κάνετε κανένα περαιτέρω σχόλιο. Όχι, σας ευχαριστώ και προσβλέπω στην επόμενη επίσκεψή μου σε εσά σε δύο περίπου μήνε. Ευχαριστώ. Nous passons maintenant au point 8 de l'ordre du jour sur les modalités, modalités de l'établissement d'un Περνούμε τώρα στο επόμενο θέμα, το οποίο είναι η δυνατότητα θέσπισης ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία. Ο εισηγητής είναι ο κύριος Σβένσον. Η υπεύθυνη επί επιτροπή είναι η ΑΦΕΤ. Ο κύριος Βένσον έχει το λόγο. Ja, det kan väl inte vara något annat än rimligt att vi i DV också ska ha Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα πρέπει να γνωμοδοτήσουμε το θέμα αυτό του Ευρωπαϊκού Ταμείου για την Δημοκρατία. το ευρωπαϊκό κληροδότημα για τη δημοκρατία. Χάρη σε εσά, κυρία Πρόεδρε, και με βάση το άρθρο 50 μπορούμε να εκφράσουμε την άποψή μας για αυτό το θέμα. Το ζήτησε αυτό η πρόεδρος, η κυρία Ζολή, αλλά μας το αρνήθηκαν, δεδομένου ότι... Είναι κρίμα όμως, διότι η Επιτροπή μας, η Επιτροπή Ανάπτυξης, γνωρίζει τι συμβαίνει όταν ε, χωλαίνει πολλές φορές η δημοκρατία η ελίπη. Πρέπει να πω ότι πρέπει η γνωμοδότησή μας να είναι πάρα πολύ συνοπτική, έτσι προβλέπετε. Και υπάρχουν τέσσερα σημεία πολύ σημαντικά όσον αφορά την δημοκρατία. Βεβαίως η δημοκρατία δεν είναι μόνο, είναι κάτι πολύ περισσότερο αν θέλετε από μια δημόσια διοίκηση και εκλογές σωστά. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να προωθήσουμε δημοκρατία και τι αξίε τη ανά τον κόσμο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να έχει κάθε ανθρώπινο όν δικαιώματα και να απολαμβάνει πλήρως από τα δικαιώματά του. Νομίζω ότι οι ελεύθερες και δίκαιες εκλογές πολλές φορές μπορούν να οδηγήσουν σε αποφάσεις που πολλές φορές δεν είναι δημοκρατικές. Υπάρχουν εδώ πάρα πολλά αμφιθελεγόμενα θέματα και θα ήθελα να σας πω ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με όλες τις ε, οργανώσεις ε, που θέλουν ε, να μαχηθούν υπέρ της δημοκρατίας και να καταπολεμήσουν τα δημοκρατικά καθεστώτα. Θα ήθελα λοιπόν όλα αυτά να λέγονται σε ορισμένε χώρες με τρόπο πιο κατανοητό και λεπτομεριακό. Ξέρω ότι υπάρχουν χώρες οι οποίες ακολούθησαν την οδό προς τον ε, εκδημοκρατισμό και θα πρέπει να θεσμοθετιστούν ε, κάποιε οργανώσεις που προασπίζονται αυτά τα δικαιώματα και να ενισχυθούν. Τρίτη παρατήρηση, θα πρέπει η αναπτυξιακή βοήθεια ή οποιαδήποτε βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι συνεχτική προς την δημοκρατία και θα πρέπει να αποφύγουμε τις επικαλύψεις. Γι' αυτό θα πρέπει ό,τι κάνουμε να το κάνουμε με τρόπο αποδοτικό, ώστε να μην υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των ε, μέσων που διαθέτουμε και να δούμε πώς θα υποφεληθούμε και από την εμπειρία που υπάρχει στον τομέα αυτό. Βεβαίως υπάρχουν κάποια πράγματα αμυγός, τεχνικά, διοικητικά ή τυπικά, αλλά νομίζω ότι η... ό,τι οτι κανουμε προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να το κάνουμε με τρόπο συμπληρωματικό και όχι ανταγωνιστικό. Σημείο 4, κυρία Πρόεδρε, για να μπορέσουμε να είμαστε αποτελεσματικοί, θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε όχι μόνο στις χώρες μας, αλλά και στις χώρες μας τις ε, ε και να παίρνουμε πάντα αποδοτικά μέτρα, διότι η έλλειψη δημοκρατίας δημιουργεί βάσανα και προβλήματα στους λαούς. Και ώρες ώρες μας μπλοκάρουν τα γεωγραφικά όρια. Θα πρέπει να ξεπεράσουμε τέτοιου δυσκολίες. Γι' αυτό η δράση μας θα πρέπει να υπερβεί τα σύνορα. Αυτά είχα να πω κυρία Πρόεδρε, συνάδελφοι, περιμένω τις παρατηρήσεις σας και βεβαίως μπορείτε να καταθέσετε τροπολογίες για τη βελτίωση του κειμένου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Συγγνώμη Πρόεδρο, δεν μπόρεσα να ακούσω τίποτε. Άκουσα το όνομά μου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Σβένσον για την έκθεσή του. Αυτό το οποίο με εκπλήσει είναι ότι αναφέρεται κάποια θέματα που αφορούν αυτό το ευρωπαϊκό κληροδότημα για τη δημοκρατία. Περί τίνος ε, πρόκειται, διότι υπάρχουν ήδη κάποιες άλλες οργανώσεις, παρατηρητήρια, με αυτά τα θέματα ασχολείται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θέλουμε τώρα... Έχουμε και ένα νέο γραφείο την πρόθεση της ε, κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Πολλά πράγματα προς αυτήν την κατεύθυνση έχουν γίνει. Δεν θέλω να πω αλλά θα ήθελα να μου πείτε Περί τίνος πρόκειται. Τι είναι αυτό το ευρωπαϊκό κληροδότημα η δημοκρατία για μας, εμάς αφορά τις ε, αναψώμενες χώρες. Και από ό,τι κατάλαβα ακόμη δεν έχει τεθεί σε λειτουργία, δεν έχει γίνει πραγματικότητα. Και τι θα λάβουμε υπόψη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα πολιτιστικά, θέματα οικονομικά, κοινωνικά, τι θα κάνουμε, θα χρηματοδοτούμε πολιτικά κόμματα. Ή θα είμαστε μακριά από πολιτικά κόμματα. Δεν ξέρω αν ε, μπορούμε να κάνουμε κάτι το κατανοητό για την έκθεση. Τέλος πάντων, πείτε μας περισσότερο περί τίνος πρόκειται. Και ποια είναι η προσθέμενη αξία κυρίως αυτού του ευρωπαϊκού κληροδοτήματος για τη δημοκρατία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ η κυρία Ντεκάιζερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Μιλήσαμε ακόμα ήδη πολύ για το κρεδότημα αυτό για τη δημοκρατία που αυτή τη στιγμή δεν είναι παρά μια ιδέα ακόμα. Γιατί νομίζω ότι ο ρόλος λοιπόν της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και δική μας είναι να ορίσουμε τι θέλουμε να είναι αυτό το κληροδόχημα. Αυτή δεν είναι τίποτα. Δεν έχει αποφασιστεί. Ποια θα είναι λοιπόν η δομή που θα δοθεί σε ποιο θα έχει επίδραση, πώ θα λειτουργήσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το πούμε αυτό, να πούμε τι θέλουμε και ιδίω να πούμε τι δεν θέλουμε. Νομίζω ότι όπως είπε ο κύριος Φένσον, η ιδέα είναι να μην έχουμε επικαλύψεις με κάποια ισχύοντα μέσα και αν το ταμείο αυτό χρηματοδοτηθεί όπως φαίνεται από τον ευρωπαϊκό προπολογισμό, εν μέρει τουλάχιστον, το Κοινοβούλιο θα διατηρήσει την αρμοδιότητά του του προσανατολισμού των πόρων αυτών και της εξέτασης ε, της χρήσης. Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποσχέσεων το κάνει, φαντάζομαι. Πρέπει να το υποθυμίσουμε όμως. Υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν έχουν αποφασιστεί και για τα οποία δεν υπάρχει συνένεση. Θα ήθελα να αναφερθώ στην παράγραφο 2, κυρία Σφένσον, όπου δικαίως λέτε και συμφωνώ μαζί σας ότι θα πρέπει να υπάρχει μια σαφής προσθέμενη εξής σχετικά με αυτό που υπάρχουν ε, αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Υπάρχει εδώ μια διαμάχη. Δηλαδή, αυτό που θα έχει την μορφή δωρεών, τα μικρά ποσά που θα έχουν σε στόχο να προωθήσουν τη δημοκρατία, θα δοθούν στους ενδιαφερόμενους των εν χωρών που αφορούνται από μια δημοκρατική μετάβαση ή πολιτικά ιδρύματα στην Ευρώπη, στην περίπτωση κατά οποία δρούν στις εν λόγω χώρες, να ωφεληθούν από τις δωρές αυτές. Στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων δεν μπορεί να δοθεί η λύση εκεί. Εγώ πιστεύω ότι αν πρόκειται για μικρά ποσά που δίνονται σε που δρούν επί τόπου, στι χώρε αυτέ που βρίσκονται σε μια φάση μετάβαση, γιατί πρέπει τα πράγματα να πάνε γλίγορα, γιατί ε, θα πρέπει ε, να τους δοθούν αμέσως γιατί δεν ε, τους χρησιμεύουν οι διάφορες ευρωπαϊκές οργανώσεις. Λοιπόν, στην περίπτωση αυτή δεν πιστεύω εγώ ότι θα μπορούμε να δώσουμε στα ευρωπαϊκά ιδρύματα που έχουν τη δυνατότητα διαχείρισης και οργάνωσης. Ακόμα και άμα πάνε στην Τινησία ή κάπου αλλού γιατί μου φαίνεται ότι αυτό θα ήταν μια στρέβλωση του αρχικού στόχου του ενόγω κληροτήματο. Να βοηθηθούν δηλαδή εκείνοι που τώρα ξεκινάνε και δεν μπορούν να βρουν μόνο τους τη λύση. Εγώ από πλευράς μου και από την ομάδα μου θεωρώ ότι τα ταμεία αυτά θα πρέπει να χρηματοδοτήσουν τις εν λόγω χώρες, το πληροδότημα αυτό μάλλον, θα πρέπει να χρηματοδοτήσουν τις εν λόγω χώρες που χρειάζονται μετάβαση προς τη δημοκρατία. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα σημείο πάρα πολύ σημαντικό. Η δυνατότητα γρήγορης δράσης στην περίπτωση αυτή είναι το σημείο που ε, δικαιολογία θέλετε αυτό το πληροδότημα Υπάρχουν όμως και κάποιες επικαλύψεις. Ήμασταν την περασμένη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη, στα Ηνωμένα Έθνη, με τον κύριο Λάμστορφ και με κάποια άλλη μέλη του Κοινοβουλίου και είδαμε το Ταμείο Εκδημοκρατισμού των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο χρηματοδοτείται από έξι τουλάχιστον από τα κράτη-μέλη. Τι θα γίνει λοιπόν, θα υπάρχει κάποιος οργανισμός μεταξύ της πρικοδότησης ε, του Ταμείου για την εκδοχημασμό των Ηνωμένων Εθνών και του ε, κληροδοτήματος του δικού μας. Και πάλι υπάρχουν αυτές οι γλίγορες ε, παρεμβάσεις, ε, όχι μεγάλης εμβέλειας κλπ. Πώς θα οργανωθούμε λοιπόν. Δεν υπάρχει μόνο επικάλυψη με τα υπάρχοντα μέσα αλλά και με κάποια μέσα που αυτή τη στιγμή χρηματοδοτούν και από τα κράτη-μέλη. Λοιπόν, καταλαβαίνω βέβαια τον στόχο του κληροδοτήματος και συμφωνώ με την ιδέα του ότι θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ χρήσιμο, αλλά θα πρέπει όμως να το καθοδηγήσουμε με μεγάλη ακρίβεια για να μην κάνουμε κάτι το οποίο θα ήταν κάτι το παραπάνω σε όλα αυτά που γίνονται για δημοκρατία και να χάσουμε κατά κάποιον τρόπο τον έλεγχο του προεπιλογισμού που θα χορηγηθεί. Αυτά και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, νομίζω ότι αυτό το σημείο είναι πολύ θετικό. Μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι ότι η ανάπτυξη των ελπισόμενων χωρών εξαρτάται βεβαίως από το επίπεδο δημοκρατίας και από την καλή διακυβέρνησή τους. Ας πούμε στην Αφρική υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν καλύτερη διακυβέρνηση και καλύτερο επίπεδο δημοκρατίας και επομένως ε, είναι σε θέση καλύτερα να χρησιμοποιήσουν την δικιά μας βοήθεια. Όσον αφορά λοιπόν την αναπτυξιακή βοήθεια, ε, ένα σημαντικό ερώτημα ε, το πολύ σημαντικό μάλιστα είναι η δυνατότητα ανάπτυξης της δημοκρατίας. Και ε, βεβαίως ε, η αποφυγή επικάλυψης είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν θέλουμε επικαλύψεις. Θέλουμε να προσπαθήσουμε να βρούμε αυτή την, αυτή την επιπλέον αξία. είναι ε, την ειδική λοιπόν προστιθέμενη αξία. Εδώ και πολλά χρόνια πολλοί οργανισμοί προσπαθούν να βελτιώσουν την ποιότητα της δημοκρατίας και της ε, σωστής διακυβέρνησης στις αναπτυσσόμενες χώρες χωρίς πολλά πολλά καλά αποτελέσματα. Ίσως δεν πρέπει να είμαστε εξαιρετικά αισιόδοξοι, αλλά εν πάση περιπτώσει ε, θα πρέπει να δούμε κατά πόσον θα πρέπει να βοηθήσουμε και τις ντόπιε οργανώσεις, γιατί υπάρχουν πολλές οργανώσεις οι οποίες μπορούν ε, να ε, έχουν την την χρηματοδότησή μας. Το σημαντικό είναι... Το σημαντικό είναι να υπάρχει ισορροπημένη εταιρική σχέση και όχι μονάχα η μία πλευρά να, κάνει, να τα κάνει όλα. Εάν πρέπει να χρηματοδοτήσουμε λοιπόν τόποιε οργανώσεις, τότε και μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό, τότε θα είναι μια πραγματική εταιρική σχέση. Και αυτό είναι πολύ σοβαρός αντικειμενικός στόχος που πρέπει να έχουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και ο κύριος Άννα Ρόλζουμ έχουν το λόγο. Ε, you, um, <coughs> Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτησή σας εδώ. Δύο λόγια έχω να πω, ενδεχομένω, ανταποκρινόμενος ε, απαντώντας μάλλον σε κάποιες από τις ερωτήσεις ε, που ε, τέθησαν σχετικά με μια αντίληψη που έχει δημιουργηθεί. Στο κοινό ανακοινωθέν 25 η Μαΐου σχετικά με τη νέα πολιτική γειτονία αναφέρθηκε και η Υπηρεσία εξωτερική Δράσης και την 20η Ιουνίου στα πλαίσια του Συμβουλίου ε, Υπουργών Εξωτερικών προωθήθηκαν κάποιες συγκεκριμένε προτάσεις. Υπήρξε μια πρόταση η οποία ξεκίνησε από τον Πολωνό Υπουργό Εξωτερικών ε, με στόχο την δημιουργία ε, ενός, μιας νέας μορφής για το ευρωπαϊκό κληροδότημα για τη δημοκρατία, κάτι σαν σύμβαση ας πούμε. Και επίσης, στα πλαίσια της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης, δημιουργήθηκε ε, μια ομάδα εργασίας ε, η οποία προσπάθησε να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο έτσι, ε, το ευρωπαϊκό κληροδότημα για τη δημοκρατία να γίνει πιο συγκεκριμένο δεν ξέρουμε πότε θα μπορέσει το κληροδότημα αυτό να αρχίσει να ε, είναι επιχειρησιακό, ε, ίσως δύο-τρία χρόνια, αλλά θα μπορούσε τελικά να πάρει τη μορφή ενός ενδιαμέσου ε, με τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις, τα κράτη-μέλη τα οποία ενδιαφέρονται να συνεισφέρουν, να, οικονομικά να το κάνουν. Και μόλις δημιουργηθεί αυτό το κληροδότημα, τότε θα ε, παίρνει χρήματα από τον ε, προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επίτροπος ε, για την Διεύρυνση ανέφερε ότι ενδεχομένως θα μπορούσαν να δοθούν σαν αρχική χρηματοδότηση 5 με 10 εκατομμύρια σε 2-3 χρόνια δηλαδή μετά την θέση λειτουργία του πληροδοτήματος υπάρχουν χώρες μεταξύ των οποίων και η Πολωνία που έχουν δείξει μεγάλο ενδιαφέρον για το θέμα. Για να σας τα πω με λίγα λόγια, ε, αυτή τη στιγμή έχει επιτευχθεί συνένεση στις υπηρεσίες και όσον αφορά ε, την, ε, το βάρος και την προστιθέμενη αξία, την οποία θα έχει το κλειοδότημα αυτό, πράγμα που αναφέρθηκε και εδώ. Ε, η αποφυγή οποιασδήποτε επικάλυψης με υφιστάμενες δομές επίσης έχει σημειωθεί και μάλιστα ορθώς ε, επεσήμαναν οι βουλευτές ότι ε, η μη επικάλυψη ε, θα δώσει τη δυνατότητα το Ευρωπαϊκό Κληροδότημα ε, να ε, δράσει, να ενεργήσει σαν μια επέκταση της δυνατότητας ανθρωπιστικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως εκεί που χρειάζεται άμεση βοήθεια, κυρίως σε χώρες που βρίσκονται σε διαδικασία δημοκρατικής μετάβασης, χωρίς όμως να έχουν ξεκινήσει ακόμα αυτή τη δημοκρατική μετάβαση actors, um, ε, και βεβαίω ε, να βοηθούμε και δημοσιογράφους και bloggers ε, και ανθρώπους που μέχρι τώρα δεν καλύπτονται από την ανθρωπιστική βοήθεια. Καταρχάς, στη, στα πλαίσια της πολιτικής γειτονίας. Να μην ξεχνάμε ότι αυτή η ιδέα προέκυψε με μεγαλύτερη ένταση μετά από την έναρξη της Αραβικής Άνοιξης Η πρότασή μας όμως ε, δεν ε, ε, είναι αποκλειστική στα πλαίσια της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης, αλλά σαν ένα από τα στοιχεία της. Επίσης μπορούν να συμμετάσχουν χώρες οι οποίες βρίσκονται εκτός πολιτικής γειτονίας. Και φυσικά θέλουμε να έχει και διευρυμένη εντολή ε, και πολλοί ομιλητές ορθώς ανέφεραν ότι η δημοκρατία δεν γνωρίζει σύνορα και αυτή είναι και η δικιά μας άποψη. Επίσης μπορούν ε, να συνεχιστούν οι συζητήσεις που έχουν ξεκινήσει με διάφορα άλλα ταμεία, με διάφορα άλλα κληροδοτήματα, έτσι ώστε να βοηθηθούν μέσω ευρωπαϊκής χρηματοδότησης ε, οι, όσοι δρούν επιτόπου και ενδεχομένως να χρηματοδοτηθούν οι δραστηριότητές τους. Αλλά η πρωτεύουσα χρηματοδοτική δραστηριότητα ε, θα αφορά αυτές τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Ε, και για μία ακόμα φορά η βοήθεια των τόπιων οργανώσεων είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Η προστιθέμενη αξία επίσης μας απασχολεί περισσότερο, ε, μας απασχολεί πολύ. Θέλουμε να μάθουμε από την γνώση τους και από τη δράση τους έτσι όπως έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Το Συμβούλιο Εξωτερικών της Παρασκευής ε, έλαβε γνώση των όσων έχουν αναλευθεί μέχρι τώρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα υπήρξε και μια δήλωση που μοιράστηκε στα κράτη-μέλη την προηγούμενη εβδομάδα ε, έτσι ώστε να την μελετήσουν και να γίνει συζήτηση με τα κράτη-μέλη ένα από τα πιο ευαίσθητα θέματα ήταν το κατά πόσον ε, θα επιτραπεί η άμεση χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων. Αυτό είναι ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα. Εμείς βέβαια δεν είχαμε σκεφτεί ότι κάποιος θα μπορούσε να κάνει επιταγή εν λευκό σε οποιαδήποτε πολιτική ομάδα, ε, πολιτικό σχηματισμό ε, και ότι άμεση χρηματοδότηση θα μπορούσε να δοθεί μονάχα σε εξαιρετικές περιπτώσεις. μελετήσαμε τον τρόπο με δράσεις άλλων οργανώσεων και προέκυψε όντως ότι μερικές φορές υπάρχει άμεση χρηματοδότηση, αλλά δεν είναι δικό δικιά μας πρόθεση ε, να έχουμε ιδεολογικά κριτήρια ή οτιδήποτε άλλο ή να στρέψουμε τη μία πολιτική ομάδα απέναντι στην άλλη. Εμείς δεν έχουμε ιδεολογικό πρόσημο. Το άλλο ζήτημα, για να ολοκληρώσω κιόλας, αφορά την ιδέα ότι το πληροδότημα θα αφορά τις ε, χώρες μέλη οι οποίες ενδιαφέρονται να συμμετέχουν οικονομικά. Κάποιες χώρες ε, προτιμούσαν ε, όλες οι χώρες μέλη να προσυπογράψουν την απόφαση. Η συμβολή του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να μελετηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, άρα αφορά ένα αργότερο στάδιο. Θα συζητηθεί πάντως το θέμα ξανά στα κράτη-μέλη. Ευελπιστούμε ότι μέχρι το τέλη τρέχοντος έτους ε, θα γίνει πιο συγκεκριμένο το ε, θέμα αυτό, η ιδέα αυτή, έτσι ώστε να γίνει ακόμη πιο συγκεκριμένο μέχρι τον, ε, την άνοιξη του 12. Πιστεύουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό όσο γίνεται πιο γρήγορα να λειτουργήσει το εργαλείο αυτό, γιατί δεν έχουμε την πολυτέλεια να περιμένουμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Αλεξάνδρ Σάντλη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Um, thank you, Madam Chair. My name is Andra Nerishanu, and I'm a miss, not Um, I don't actually, I work in... Αλεξάνδρα και όχι η Alexander... Δεν έχω να προσθέσω και πολλά στα όσα είπε ο συνάδελφος από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Υπάρχει συνένεση ε, μεταξύ ε, της, Επιτροπή, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης σχετικά με όλα αυτά τα οποία ανέφερε. Και υπάρχει εκφρασμένη βούληση, ας την πούμε έτσι, για τη δημιουργία του κληροδοτήματος αυτού. Αλλά βεβαίως θα πρέπει πρώτα να δημιουργηθεί η δομή πριν αρχίσει κανείς να συμβάλλει στο κληροδότημα αυτό. Ε, και Βεβαίω, θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η οποιαδήποτε χρηματοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό μέσω του κληροδοτήματος θα γίνεται με συγκεκριμένο τρόπο και υπό συγκεκριμένες προποθέσει και με τρόπο ώστε να συμβάλλει στην προστιθέμενη αξία του κληροδοτήματος ε, που θα αφορά κυρίως την εξέβρεση συμβεστικών λύσεων σε ε, περιπτώσεις χωρών που βρίσκονται ε, στη διαδικασία εκδημοκρατισμού. Θα υπάρχουν συμβολές και από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό και από τον Προϋπολογισμό των κρατών μελών, αλλά ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι κανόνες ε, είτε της χρηματοδότησης είτε της πρόθεσης της χρηματοδότησης. Ε, για να ολοκληρώσω να πω ότι θέλουμε, προσδοκούμε την ολοκλήρωση των ε, συζητήσεων μεταξύ της Κομισιόν και του, των χωρών μελών, έτσι ώστε να υλοποιηθεί το κληροδότημα αυτό. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Θα το Ο κύριος θα έχει το λόγο για να ολοκληρώσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Προσβλέπω πραγματικά στις ε, προτινόμενες τροπολογίες. Ε, Βέβαια, υπάρχουν ε, κάποιες επικαλύψεις, Πρόεδρε, αλλά ο κίνδυνος είναι ότι ίσως τελικά μιλάμε για δημοκρατικές αξίες χωρίς να αναλύσουμε τι εννοούμε και τι ακριβώς θέλουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό νομίζω, όχι μόνο εδώ, γενικά. Να σκεφτούμε εις βάθος τι εννοούμε όταν λέμε δημοκρατία, ποιες είναι οι αξίες τις οποίες αναφερόμαστε. Ίσως οι αξίες είναι εκείνες που μας προσφέρουν τη δημοκρατία και όχι τα είναι πάρα πολύ επίγον λοιπόν να έχουμε καλύτερη εικόνα του τι συζητάμε. Αυτή η όρη θα πρέπει να είναι ξεκάθαροι. Μπορούμε να εργαστούμε στην Αφρική, αλλά όχι μόνο στην Αφρική βέβαια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε αυτή τη συζήτηση για δημοκρατία, δημοκρατικές αρχές, για ανθρώπινα δικαιώματα, Πρέπει λοιπόν να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση. σα. ευχαριστώ λοιπόν για όλες τις προτάσεις και τις ιδέες που προσφέρετε, πρόεδρο. Ευχαριστώ. Σας υπενθυμίσω ότι 8 Δεκεμβρίου μεσημέρι είναι η προθεσμία για την υποβολή ε, και η ψηφοφορία θα γίνει στις 25 Ιανουαρίου. Τώρα θα περάσουμε στην ψηφοφορία. Σας παρακαλώ πάρτε τις κάρτες σας στο χέρι.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 Donc tout le monde a sa la boîte euh, ad hoc. Λοιπόν, θα ψηφίσουμε το σημείο 9. Αλλά κάνουμε ένα τεστ πρώτα. Άκρη ψηφοφορία.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 La politique étrangère de l'Union européenne à l'égard des η εξωτερική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι των χωρών B και άλλων αντιωμένων δυνάμεων. Στόχοι και στρατηγικέ. Συμβαστική 1. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Κατά τμήματα ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχή. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Mm. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Α, να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Le vote est clos. Ψήφισαν όλοι. Α, ναι, απερίφθη. Τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 13 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 2. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 19. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 20. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 22. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Α, τελική ψηφοφορία. Α, μάλιστα. Ωραία. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία άρχεται. Encore une voix qui manque. vote est clos. Adopté l'unanimité. Ομόφωνα να κρυθεί. Ωραία. Σημείο 10 σήμερα τη διάταξη. Πρωτόκολλο που συμφωνήθηκε μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Δημοκρατία τη Γουινέα Βυσσάου σχετικά με τον καθορισμό ελευτικών δυνατοτήτων. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. ηλεκτρονικό ψηφοφορία για το, το τέλος, για να εγκρίνουμε την ε, πρόταση αυτή της γραμματότησης. Ολοκληρώθηκε ομόφωνη έγκριση. point 11 à l'ordre des jours. La... σημείο 11 Αναπτυξιακή συνεργασία τη Ευρωπαϊκή Ένωση και Καθολική Καθολικής στην Ενέργεια στο 2020. Τροπολογία 14, ε, 30 με συγχωρείτε. Υπέρ, κατά. Αποχέ, εγκρίνεται. 15. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 16. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 17. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 18. Χωριστή ψηφοφορία. Ψηφίζουν το πρώτο μέρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το δεύτερο υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Όχι. Απορρίπτεται. Ηλεκτρονική επελίδευση Για το δεύτερο μέρος. Έληξε ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Μ' 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 20. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 21. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 22. Προφορική τροπολογία. Υπέρ, κατά, αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση της 22 αρχίζει η ψηφοφορία λίγη ψηφοφορία εγκρίθηκε «23 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται». 24 υπέρ καλά, κατά αποχές εγκρίνεται 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 26 κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 27 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. <coughs> Ηλεκτρονική επαλήθευση. Αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 29. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 30 <clears throat> υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 31 και 32 αποσύρονται, 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 34. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 35. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 36. προφορική τροπολογία πάλι, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 37. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 38. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 39. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία 43. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πίπτη 43, περνάμε στη 44, υπέρ. Ψηφίζουμε χωριστά. Αρχίζουμε με την ψηφίση του πρώτου μέρους. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται το πρώτο. Qui est Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 46. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 47. Προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται όχι ηλεκτρονική επαλήθευση αρχίζει η ψηφοφορία η... Λίγη πληροφορία και απορρίπτεται η τροπολογία. 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 52 υπέρ Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ή 53. Έχει αποσυρθεί το αρχικό κείμενο της παραγράφου 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται.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 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 1. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 2. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 3. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Θα ψηφίσουμε τώρα το σχέδιο έκθεσης έτσι όπως τροποποιήθηκε. Αυτή η ψηφοφορία Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίθηκε η έκθεση με 17 προς 3 ψήφους. Fin 12 de l'ordre du jour européenne et la Chine. Ε, σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Κίνας. Συμβιβασμός ε, Β. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβασμός C. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Τι να σας πω. Μάλλον θα ε, ε, κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση. Συμβιβασμός σε. Άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία λοιπόν. Λείπει μία ψήφος.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 Τροπολογία 26 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 27 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 29 κατά τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Διαμαρτυρίες, επαλήθευση δεύτερο τμήματος τροπολογίας 29, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Κατά δύο ψήφους. Συμβιβασμός D. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Όχι. Εγκρίνεται. Εντάξει, ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται, είπαμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 33. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 34. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 35. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 36. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός Ι, κατά τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Διαμαρτυρίες. Επαληθεύουμε λοιπόν, επαλήθευση ηλεκτρονική, άρχιτη ψηφοφορία για το δεύτερο τμήμα. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με δύο ψήφους διαφορά. Εγκρίθηκε λοιπόν αυτό. Περνάμε στην τροπολογία 41. Υπέρ. Τροπολογία 41 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία 2 Λοιπόν, μαθαίνω ότι η προφορική τροπολογία υπαριθμών 2 έχει ήδη αποσυρθεί, επομένως περνάμε στην τροπολογία 45. Έχει ζητηθεί ψηφοφορία κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα λοιπόν στην τροπολογία 45 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 45 υπέρ κατά αποχές Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει ηλεκτρονική υπαλήθευση. Δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 45 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 47. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τραπολογία 48 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 50 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβασμός F. Κατά τμήματα η ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Εγκρίνεται, συγγνώμη, λέει η Πρόεδρος. Εγκρίνεται. Περνάμε επομένως στην τροπολογία 57. Τροπολογία 57 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 59 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 61 κατά τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Τροπολογία 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται.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 κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές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 ψήφισαν όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας και εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. avec On Nous passons maintenant Ολοκληρώσαμε λοιπόν ε, τις ε, ψηφοφορίες και περνάμε τώρα στην γνωμοδότηση για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Συγγραφεύς ε, της γνωμοδότησης αυτής είναι ο κύριος Μπαρτ Στάς. Ε, αφορά την δράση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, κυρίως όσον αφορά την ανάπτυξη και θα του δώσω το λόγο αμέσως. Και μετά θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ε, για πέντε το πολύ λεπτά. Τον λόγο έχει ο κύριος Μπαρτ Στάσ Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ehm, eh, Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Η γνωμοδότησή μου ήταν πάντα πολύ σύντομη. Αυτό έπρεπε να κάνω κιόλα. Έπρεπε να περιοριστώ σε πολύ συγκεκριμένο αριθμό παραγράφων. Ε, βέβαια συνεργάστηκα και με τους χιλιάδες εισηγητές. Εκ των υστέρων Πάντα μπορεί κανένας να παρατείνει την έκθεση με τροπολογίες που θα τύχουν συνένεσης. Οπότε θα είναι πολύ πιο ισχυρή, αν θέλετε, η γνωμοδότηση αυτή στο περιεχόμενο σας. Ξέρετε, το έργο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεις ασχολείται με διάφορα σχέδια στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, εξωτερικά στοιχεία είναι μάλλον περιορισμένα, δηλαδή η μαγιά είναι 90 προς 10. Παρ' όλα αυτά, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει μεγάλη δυνατότητα επίδρασης στους εταίρους μας ε, στις αναπτυσσόμενες χώρες. Εγώ διατύπωσα 7 προτάσεις, ξεκινώντας από την απόφαση που δημιουργήθηκε φέτος το Σεπτέμβριο. Πρόκειται για εγγυήσει ε, για απώλειες της ΕΤΕΠ ε, από κάποιες επενδύσεις. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο γιατί αν κοιτάξουμε την ε, έκθεση βλέπουμε ότι οι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί είναι πάρα πολύ καλοί. Καλύτεροι από ό,τι περίμενα ομολογώ. Αλλά αυτά η γενική μου σύσταση παραμένει. Ότι δηλαδή θα πρέπει εμείς σαν κοινοβούλιο θα πρέπει να υποβάλουμε ερωτήσεις όσον αφορά τις πρωτοβουλίες της ΕΤΕΠ όπου θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη ότι οι πρωτοβουλίες αυτές θα πρέπει να είναι απόλυτα σύμφωνες με τη συνθήκη. Η συνθήκη της αγώνας είναι πάρα πολύ αναλυτική. Ξέρουμε ότι αποτελεί ένα, μια πολύ καλή βάση και αυτό θέλω αυτή η διατύπωση να παραμείνει ως έχει. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ήρθε σε διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδίω με την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού τελευταία και υπάρχουν πάρα πολλά θετικά στοιχεία. Εγώ παραδείγματο χάρη αναφέρομαι ρητά στο δεύτερο σημείο στις ε, κλιματικές αλλαγές. Γιατί ξέρουμε βέβαια ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες είναι εκείνες που πλήττονται περισσότερο από τις επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών. Και θα είναι καλό να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας και να βοηθήσουμε τις ε, χώρες αυτές. Επίσης, ε, αν το παρουσιάσουμε αυτό στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεως νομίζω θα αντιδράσει δηλαδή ότι τα έργα για την τροφοδότηση με ενέργεια θα πρέπει να είναι μικρής κλίμακας. Υπάρχουν βέβαια και μεγάλα σχέδια υποδομών που καμιά φορά έχουν και αρνητικές επιπτώσει. Αυτό είναι κάτι που ε, οδηγεί και σε πολλή αντίδραση στον, ε, στα ΜΜΕ. Λοιπόν, θα πρέπει να συγκεντρώσουμε την προσοχή, νομίζω δηλαδή ότι συγκεντρώνεται ιδιαίτερη προσοχή στα, ε, στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο. Επίσης ε, λέγεται ότι θα πρέπει και οι οικολογικέ και κοινωνικές πτυχέ τη πολιτική να λαμβάνονται περισσότερο υπόψη που δεν γίνεται αυτή τη στιγμή στις τρίτε χώρες και γι' αυτό συστήνω στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να, επιδώσει περισσότερη σημασία στο σημείο αυτό. Μια άλλη πρόταση. Ας προσπαθήσει να συνδέσει τα διάφορα μέσα ε, της παραδείγματο χάνει για την επίτευξη των στόχων της χιλιετίας ή για την καταπολέμηση της φτώχειας βέβαια συμπεριλαμβανομένου και του σεβασμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίσης να λαμβάνουν υπόψη και κάποια σχέδια που έχουν περισσότερη ε, κοινωνική ε, απόδοση. Επίσης θα πρέπει να δοθεί η μεγαλύτερη σημασία στις οικολογικές αρχές. Καλό τέλος να, ζητήσει, να λάβει υπόψη πολύ περισσότερο τις κοινωνικές πτυχές η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σε όλα τα στάδια των σχεδίων. en voltooid wordt om daar... Uh... Δηλαδή όχι μόνο στην αρχή αλλά και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και ολοκλήρωσης των σχεδίων αυτών. Και επίσης οι διάφοροι δείκτες επίδοσης θα μπορούν να καταδεικνύουν κατά πόσο τα πράγματα λειτουργούν σωστά ή όχι. Και γι' αυτό θα πρέπει να είναι πιο ακριβής άλλη πρόταση, κάτι που γίνεται ήδη ότι δηλαδή χρειάζομαι καλύτερη παρακολούθηση των συνολικών δανείων που δίνονται, δηλαδή και εκείνο που δίνονται στις ε, ΜΜΕ θα πρέπει να εξετάσετε κατά πόσον επιτυχάνουν τους στόχους τους και θα πρέπει να υπάρχει επίσης μεγαλύτερη διαφάνεια και η λογοδοσία να είναι πολύ καλύτερη. Και τέλος, θα πρέπει να υπάρχει περισσότερη οικολογική αηφορία. Και τέλος, θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεως να τηρεί πάντα τους κανόνες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι κάτι που απορρέει από την συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά πρέπει να τηρούμε και διεθνή πρότυπα, οικολογικό τομέα, κοινωνικό τομέα. Αυτό θα πρέπει να είναι η συστηματική προϋπόθεση όσον αφορά την πρόσβαση των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τραπεζα Επενδύσεων. Και τέλος θα ήθελα να προτείνω ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες εργάζονται κατά αυτών των προτείνων, των προτύπων συγγνώμη, θα πρέπει να εγγραφούν σε κάποιο μαύρο κατάλογο. Ένα μαύρο κατάλογο δηλαδή όπου θα αναφέρονται όλες οι επιχειρήσεις που δεν θα δικαιούνται χρηματοδόση από την ΕΤΕΠ. Και τέλος κυρία Πρόεδρε και για τη δική σας ε, πρόταση. Θα ήθελα να πω ότι εκείνες οι επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους σε φορολογικούς παραδείσους θα πρέπει επίσης να εξαιρούνται από αυτή τη χρηματοδότηση. Θα ήθελα, σε συμφωνία με τους και όλους να υποβάλω και άλλες ε, τροπολογίες. Η μία από αυτές θα είναι ότι η επίδραση τη Ευρωπαϊκή Τράπεζας θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται πολύ καλύτερα και αριθμητικά. Η αιτήσια έκθεση είναι πάρα πολύ όμορφη, αν θέλετε μπορώ να το πω έτσι. 72 δισεκατομμύρια δάνεια που δίνονται από την τράπεζα αυτή. Αυτά θα πρέπει νομίζω να είναι όμως πολύ πιο συγκεκριμένα τα στοιχεία και να αναφέρουν και οι τρίτες χώρες που παίρνουν τα χρήματα αυτά και τέλος στενότερη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής ε, Τράπεζας Επενδύσεων και των τοπικών ε, επιχειρήσεων. Και τέλος, να μην ξεχνάτε και το μνημόνιο συνεννόησης που υπάρχει ακριβώς μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων όπου λέγεται ότι θα πρέπει να συμμετάσχει πιο έντονα και εις βάθος το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από ό,τι μέχρι τώρα, όσον αφορά και την πλατφόρμα συνεργασία και ανάπτυξη. Αυτό θα μπορούμε να το αναφέρουμε συγκεκριμένα. Υπάρχει και μια πρόταση κειμένου που έχουμε μπροστά μας και που μπορούμε νομίζω να εκμεταλλευτούμε το ώστε σε διάλογο με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να φροντίσουμε να λαμβάνουμε περισσότερο υπόψη τα δάνεια αυτά ούτω ώστε να αφαιρεθούν περισσότεροι εταίροι μα ε, για τον τρίτο κόσμο. Αυτά πολύ γρήγορα εισαγωγικά. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Στάση. Το λόγο τώρα έχει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που εκπροσωπεί ο κύριος Καράνο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ κύριε Στάση για την προσπάθεια που καταβάλλετε και την καλή δουλειά που επιτελέσετε στα πλαίσια αυτής της έκθεσης. Κάποιες παρατηρήσεις σε αυτό το στάδιο από εμά. Χαιρετίζουμε πρώτα απ' όλα την συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα την Επιτροπή σα όσον αφορά τι δραστηριότητε μα εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση, που όπω γνωρίζετε και όπω ανέφερε και ο εισηγητής είναι στόχος ε, μεσοπαθμής αναθεώρησης, τα πλαίσια των αποφάσεων που έχουμε μέσω πρόθεσμα και πράγμα που αποτελεί αντικείμενο τη δική σα συναπόφαση και θα ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο. Επίση, θα πρέπει να πω ότι εδώ καλύπτεται και οι χώρε και ε, στα πλαίσια τη συμφωνία Κοτονού και είμαστε ανοιχτοί για να μοιραστούμε με εσά όλε τι πληροφορίε που έχουμε όσον αφορά αυτέ τι δραστηριότητε. Κάθε χρόνο παρέχουμε τέτοιε πληροφορίε και την επόμενη φορά στι 26 Ιανουαρίου θα γίνει η παρουσίαση του μέσου επενδύσεων μας στα πλαίσια της απαλλαγής IDF στην Ισιατική Επιτροπή, την Επιτροπή Κόμμα, όσον αφορά τώρα τις διάφορες υποδείξει του εισηγητού. Πρέπει να πω ότι τις καλωσορίζουμε. Και αυτά είναι ενθάρρυνση ώστε να βελτιωθούν τα πράγματα και να μπορέσουμε να δώσουμε ε, κάτι καλύτερο στα πλαίσια του κύριου στόχου μας που είναι η εξωτερική μας πολιτική. Απ' την άλλη θα πρέπει να λάβουμε υπόψη κάποιους περιορισμούς που αντιμετωπίζουμε σε σχέση με το επιχειρησιακό πρότυπο που ακολουθούμε και βασίζεται στο ότι είμαστε η τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπηρεσία των κρατών μελών και ο κύριος στόχος μας είναι η κοινωνική και η ε, οικονομική ανάπτυξη των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το πρότυπο λοιπόν προσπαθούμε να το προσαρμόσουμε και να το εφαρμόσουμε και εκτός ορίων Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν όμως και όρια στο τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε διασφαρίζοντας ε, και τον κύριο στόχο των δραστηριοτήτων μας. Εμείς στα πλαίσια των ε, στόχων μας έχουμε να καλύψουμε το προσωπικό, την διακυβέρνηση, το τοπικό προσωπικό, την δυνατότητα ανάληψης κινδύνων και την πρόσβαση σε κοινοτικά κονδύλια και δάνεια ενεργούμε πολύ διαφορετικά πολλέ φορέ από άλλε πολυμερεί ή διμερεί αναπτυξιακέ τράπεζες. Αυτά είναι λοιπόν τα πλαίσια με τα οποία κινούμεθα και ενεργούμε. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε σε ποιο μέτρο μπορούμε να συνεισφέρουμε στην ε, ε, αναπτυξιακούς στόχους πιο άμεσα. Δεδομένου ότι η δική μας η πρόσβαση μπορεί να και ενέργεια, μπορούμε να είναι έμεση δεδομένου ότι έχουμε περιορισμένα κονδύλια και δεν έχουμε και την δυνατότητα να αναλάβουμε κινδύνους. Πιστεύουμε ότι βεβαίως είναι στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των αναπτυσσόμενων χαλών πολύτιμος ρόλος μας, αλλά θα πρέπει οτιδήποτε θέλουν να αναλάβουν περαιτέρω να το συζητήσουμε πρώτα απ' όλα με τα κράτη-μέλη. Και ιδιαίτερος για την προοπτική του 2013, το βήμα που ανέφερε ο η είναι το πλαίσιο συζητήσεων όπου με τα κράτη-μέλη το Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο που είναι παρατηρητής και τα κράτη-μέλη μπορούμε να σκεφτούμε με ποιους τρόπους μπορούμε να ενώσουμε τις δράσεις ώστε να είμαστε πιο αποδοτικοί στις δράσεις μας. Και βεβαίως συμφωνούμε με το τελευταίο σημείο σας ότι θα πρέπει και σε αυτό το πλαίσιο να προωθήσουμε τα κοινοτικά πρότυπα. Πιστεύω ότι ό,τι κάνουμε θα πρέπει ως Ευρωπαϊκή Ένωση να το κάνουμε με τρόπο συνεκτικό και εμείς και όλα τα άλλα ε, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία συμμετέχουν σε αυτή την αυτοβήμα, σε αυτή την πλατφόρμα. Θα πρέπει λοιπόν να κινούμε από τις ίδιες αρχές ώστε να μπορέσουμε να αυξήσουμε και την, πολιτική μας, την επιρροή μας στο θέμα της πολιτικής την οποία ασκούμε. Εμείς είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε υπόδειξη εκ μέρους ώστε να μπορέσουμε να ενισχύσουμε και να διαρθρώσουμε περαιτέρω τον διάλογο και τη συνεργασία μαζί σας, Πρόεδρος. Στις 19 Δεκεμβρίου, στα πλαίσια αυτής της ετήσιας έκθεσης, ε, θα ε, παραστεί στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα έχουμε τον νέο πρόεδρό μας για αυτό το θέμα, τον Ιω Χόιερ και αν θέλετε τους επόμενους μήνες μπορείτε να τον καλέσετε να παραστεί στις εργασίες της Επιτροπής σας. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ. Η Κομισιό. Η κυρία Μέτε Πάνιγκε. αντικαθιστώ εγώ την ε, κυρία Μετεπάνενα. Ε, θα ήθελα να πω ότι καλωσορίζουμε τις ε, προτάσεις σας γιατί ευθυγραμμίζονται και με την θέση που έχουμε πάρει και τα αναφέρουμε άλλωστε και στην ενδιάμεση αξιολόγηση της εξωτερικής δράσης της τράπεζας, κυρίως για τους στόχους σχετικά με τη μείωση της ένδυας και την ανάπτυξη, την εστίαση βεβαίως και στις κλιματικές αλλαγές. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι εμείς έχουμε πάρει αυστηρή θέση όσον αφορά τα θέματα της φόρο αποφυγής και φοροδιαφυγής, καθώς επίσης και το θέμα των φορολογικών παραδείσων. Βεβαίως στηρίζομαι και το Κοινοβούλιο στην ενθάρρυνση της ε, Κεντρικής ε, Τράπεζας ε, να ελέγχει καλύτερα τις δράσεις της και όχι μονάχα αυτές οι οποίες σχετίζονται με την οικονομική απόδοση των επενδύσεων αλλά κυρίως και στο κατά πόσον προσδίδουν τη θέμενη αξία. Ο διάλογος μεταξύ των θεσμικών οργάνων που έχει ξεκινήσει μας βρίσκει απολύτω σύμφωνος και αυτά θέλαμε να πούμε. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Στάς για να ολοκληρώσει. Λοιπόν, δεν έχω ακόμα εξάγει συμπεράσματα που μπορώ να εξάγω αυτή τη στιγμή. Όμως με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολούθησα τις τοποθετήσεις των ομιλητών και υπενθυμίζω ότι είμαι και μέλος και της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού ε, μάλιστα είμαι και αντιπρόεδρος, γνωρίζω ότι ε, στην αρχή υπήρχε κάποια δυσκολία στη σχέση μεταξύ της ε, ΕΤΕ και του Κοινοβουλίου. Αυτή η δυσκολία τώρα έχει εξαλειφθεί και χαίρομαι που η θέση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας ήταν σαφής και ότι ε, ετέθη ευνοϊκά σε σχέση θετικά, σε σχέση με την πρώτη πρόταση που έκανε. Ελπίζω ότι και με τον νέο πρόεδρο ε, η συνεργασία θα είναι καλή και ότι ε, θα φέρθηκε μια νέα πνοή με τον νέο πρόεδρο. Τα θέματα τα οποία συζητάει η Επιτροπή Ανάπτυξης είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ε, και επομένως ε, με τη διπλή μου κασκέτα και σαν μέλος της Επιτροπής Ανάπτυξης και του Ελέγχου του Προϋπολογισμού θα προσπαθήσω να αντιμετωπίσω όσο γίνεται πιο σφαιρικά και συνολικά το ζήτημα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Θα περιμένουμε βεβαίως ε, και την παρουσία ΣΥ του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας από τον Πρόεδρό της ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Να υπενθυμίσω ότι 25 Ιανουαρίου του 2012 στις 11 το πρωί ε, εκπνέει η προθεσμία υποβολή τροπολογιών για την έκθεση του κυρίου Στάς, ενώ η ψηφοφορία θα λάβει χώρα στις 9 Φεβρουαρίου. Υπό τα διάφορα δεν έχουμε τίποτα. Επομένω, τελευταίο σημείο τη ημερησία διάταξη, η επόμενη συνεδρίασή μας, 8 Δεκεμβρίου 2011, δηλαδή μεθαύριο την Πέμπτη, 9 με 12.30. Θα συνεχίσουμε τώρα και κλεισμένων των θυρών ε, με την συνεδρίαση των συντονιστών. Μπορούν να είναι παρόντες μονάχα οι βουλευτές, οι βοηθοί τους, ε, το προσωπικό των πολιτικών ομάδων, καθώς επίσης ε, και οι υπάλληλοι της ε, Γραμματείας του Κοινοβουλίου. Καλό λοιπόν όλους τους ε, υπολείπους να εγκαταλείψουν την αίθουσα, να συνεχίσουν τις συζητήσεις τους εκτός ε, της αιθούσης, έτσι ώστε και εμείς να συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Σας ευχαριστώ πολύ.